I think we can start. Να ξεκινήσουμε, παρακαλώ. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer. Σας καλωσορίζω στην ακρόαση μας για το ε, για τον ε, ενιαίο χώρο ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχετε το ε, πρόγραμμα να καλωσορίσουμε και τους ε, ομιλητές μας στο Κοινοβούλιο. Ξέρουμε τα ε, όρια που έχουμε, τα χρονικά. Έχουμε πρώτα τον κύριο Ρίτσαρτ Κιούρντεν, για 10 λεπτά. Θα μας παρουσιάσει τη μελέτη για τον αντίκτυπο των αυτοκινήτων όγκου υψηλού ή χαμηλότερου όγκου και υψηλού ή χαμηλότερου βάρους για την οδική ασφάλεια, κυρίως για τους ευαίσθητους χρήστες. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Ο τίτλος της παρουσίασής μου είναι στην οθόνη σας, τον βλέπετε. Ο στόχος του project ήταν να δούμε ποιος είναι ο αντίκτυπος αν δούμε περισσότερα SUV και πολυμορφικά αυτοκίνητα στους οχήματα στους δρόμους και πώς αυτά επηρεάζουν την οδική ασφάλεια. Θα αναφέρω και κάποια ερωτήματα της ε, έρευνας. Αν τα SUV και τα πολυμορφικά είναι πιο επιθετικά σε σχέση με τα επιβατικά αυτοκίνητα, τα πιο μικρά αυτοκίνητα, κυρίως ό,τι αφορά τους ε, πεζούς και τους ε, ποδηλάτες. Δεύτερο ερώτημα αν υπάρχουν ε, ε, μειονεκτήματα στο να είναι κανείς σε ένα μικρότερο αυτοκίνητο ε, όταν βρίσκεται σε κάποιο δυστύχημα. Η έρευνα αυτή χρονολογείται εδώ και 15 χρόνια. Βλέπουμε σταθερή μείωση των θανάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, των θανατηφόρων δυστυχημάτων. Βεβαίω βλέπουμε μια σταθερή πορεία στην μείωση των θανατηφόρων δυστυχημάτων και αν δούμε από πού προέρχονται αυτά τα ατυχήματα, είναι κυρίως από επιβατικά αυτοκίνητα. Δεν είναι πολύ καλή η πρόοδος αν δούμε τους ε, ποδηλάτες, ε, τους ευαίσθητους ε, πολίτες και τους πεζούς. Λίγο background τώρα, λίγα ιστορικά στοιχεία. Έχουμε κάποιες τάσεις που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γυράσκει ο πληθυσμό της, που είναι καλό ε, άλλο ένα καλό είναι ότι οι, οι πολίτες περπατούν περισσότερο, χρησιμοποιούν πολύ περισσότερο ποδήλατα και αυτό είναι καλό, είναι και πιο υγιές. Ε, βλέπουμε ότι έχει αλλάξει και ο στόλος των οχημάτων. Βλέπουμε λιγότερο μεσαίου μεγέθους, ε, λιγότερα μεσαίου μεγέθους ε, ε, αυτοκίνητα και περισσότερα αυτοκίνητα πόλης. Έχει αλλάξει λοιπόν η αναλογία. Και επίσης βλέπουμε πολλές τεχνολογίες οχημάτων, πολλά συστήματα δηλαδή, που αναλαμβάνουν ε, την ε, οδήγηση, ας πούμε, βοηθούν την πέληση, βοηθούν το παρκάρισμα και άλλου είδους συστήματα. Αυτό λοιπόν που θα μπορούσε να προκύψει από αυτές τις αλλαγές είναι ότι θα είναι λιγότεροι οι ε, εμπλεκόμενοι σε τέτοια δυστυχήματα με μεγάλα και πολυμορφικά αυτοκίνητα. Βλέπουμε, πρέπει βέβαια να δούμε τι συμβαίνει και με τα μικρά αυτοκίνητα όταν αυτά βρίσκονται σε ατυχήματα με μεγαλύτερα οχήματα. Δεν θέλω να μιλήσω για τους κανόνες που υπάρχουν σε λεπτομέρειες. Θα μιλήσω κυρίως για τις συστάσεις μας σε σχέση με αυτούς τους κανόνες που υπάρχουν και πώς αυτοί μπορούν να βελτιωθούν. Πάμε λοιπόν στην πρώτη, στην πρώτη ερώτηση της έρευνάς μας. Αν τα SUV και τα πολυμορφικά είναι πιο επιθετικά από ένα μικρό αυτοκίνητο. Αυτό που γίνεται εδώ και πολλά χρόνια είναι ότι οι μηχανικοί μελετούν το πώς μπορεί κανείς ε, να τεστάρει τα αυτοκίνητα και να τα, καταστήσει, να τα καταστήσει πιο ασφαλή όταν χτυπήσουν έναν πεζό. Αν, ανάλογα με το αν το χτυπήσουν στο, στη λεκάνη, στο κεφάλι ή στο χέρι. Βεβαίως με τις κούκλες αυτές δεν μπορεί κανείς να έχει αξιόπιστα αποτελέσματα. Οπότε χρησιμοποιούνται ε, συγκεκριμένα, συγκεκριμένα μοντέλα τα οποία έχουμε, αναπαριστούν ουσιαστικά το, τα πόδια, την μέση και τον κορμό του, ε, του πεζού. Και ανάλογα με το που χτυπά αυτό το αυτοκίνητο καταγράφουμε τα αποτελέσματα. Η κόκκινη γραμμή που βλέπετε εδώ στη διαφάνεια αντικατοπτρίζει ένα αυτοκίνητο πολυμορφικό και βλέπετε πού θα, που θα χτυπήσει το κεφάλι του πεζού αν τον χτυπήσει. Αν βάλουμε ένα αυτοκίνητο 4x4 ή ένα SUV, πάλι αλλάζει το σημείο στο οποίο θα χτυπήσει και το, το κεφαλαίο κορμός του πεζού. Και βλέπουμε λοιπόν ε, πως, ε, ότι η μεγαλύτερη ζημιά γίνεται, προκαλείται στον ε, κορμό στη λεκάνη. Βλέπουμε ότι στο καπό του αυτοκινήτου χτυπά το, το κεφάλι του πεζού και σε ένα σεντάν ας πούμε, αυτοκίνητο θα χτυπούσε πιο χαμηλά. αν είναι πολυμορφικό πάλι ή επιβατικό πάλι είναι διαφορετικό το σημείο. Ε, βέβαια ένα μικρό κομμάτι του καπο μπορεί να ε, δοκιμαστεί. Οι κατασκευαστέ λοιπόν ε, δαπανούν πολύ χρόνο και πολύ κόπο για να σχεδιάσουν ακριβώ αυτό το κομμάτι του αυτοκινήτου ώστε να μπορεί να περάσει το αυτοκίνητο. Βεβαίω να περάσει το αυτοκίνητο στη δοκιμασία. Κάτι που μπορεί στην πράξη να μην συμβεί. Τώρα, Έχουμε συμπεριλάβει και μία μελέτη στην οποία πήρα μέρος πριν από λίγα χρόνια. Μελετήσαμε 34 ε, δυστυχήματα. Ε, μελετήσαμε κάποιου αστυνομικού φακέλους για να δούμε πού προκλήθηκαν οι, περισσότερες, ε, οι περισσότεροι τραυματισμοί και βρήκαμε την αιτία του, ε, του τραυματισμού, αν προκλήθηκε δηλαδή από το καπό ή από, τον, από τους προφυλακτήρες ή από κάποιο άλλο σημείο του αυτοκινήτου. Κανένα από αυτά τα ε, τραύματα, ε, τα σοβαρά τραύματα, θανατηφόρα ίσως, κανένα από αυτά που μελετήσαμε, από το βήμα τουλάχιστον που είδαμε, δεν ε, προέκυψε από το καπό ή από, τον, από το κομμάτι του αυτοκινήτου που θα είχε δοκιμαστεί από τον κανόνα 78, από τον οποίο περνούν τα οχήματα. Ένα επτάχρονο παιδάκι μόνο χτυπήθηκε από, το, από, το, από τον προφυλακτήρα του αυτοκινήτου και είχαμε 12 χτυπήματα στην ε, ε, Μπαρμπρίς. Για τα δυστυχήματα από χτύπημα στο κεφάλι, ε, τα περισσότερα ήταν από σημεία τα οποία δεν τεστάρονται και δεν ήταν μέσα στο πλαίσιο της έρευνας του κανόνα 78. Είναι ε, αρκετά επιτυχής λοιπόν ο ε, κανόνας. Όταν κάποιος χτυπάει στο καπό του αυτοκίνητου δεν είναι θανατηφόρα το, θανατηφόρος ο τραυματισμός. Αλλά όταν κάποιος, ε, η θανατηφόρα, τα θανατηφόρα ατυχήματα δεν προκύπτουν από το καπό του αυτοκινήτου, από χτύπημα από το καπό του αυτοκινήτου. Επίσης, οι ποδηλάτες ξέρουμε ότι είναι πολύ πιο εύκολο να χτυπήσουν, με το, να τον παρμπρί του αυτοκινήτου ή στον καθρέφτη. Και αυτό το ξέρουμε, γιατί όπως ε, όσο γυράς και ο πληθυσμός, ε, τόσο αλλάζουν και, τα, και το, τα σημεία στα οποία χτυπάει περισσότερο. Οι μεγαλύτερες μας ηλικίε χτυπούν περισσότερο στη λεκάνη ή στα πόδια. Αυτό, ε, κάτι άλλο σημαντικό επίσης είναι η ταχύτητα. Ε, η μείωση της ταχύτητας ε, είναι ακριβώς ο παράγοντας που μειώνει πάρα πολύ τον κίνδυνο θανατηφόρου στοιχήματος. Οι πεζοί κυρίω ή οι ποδηλάτες ε, πραγματικά υπόκεινται πολύ σε, τέτοιες, σε τέτοια χτυπήματα και η μείωση της ταχύτητας είναι ο αποφασιστικός παράγοντας. Αν δούμε τώρα λίγο και τη βιβλιογραφία, στην, στη ΣΥΠΑ είδαμε πολύ καλά αποδοκτικά στοιχεία, περίπου αύξηση 30% στον, κίνδυνο των θανάτου των πεζών αν χτυπηθούν από SUV. Βεβαίω τη είπα, δεν υπάρχει κανένα κανόνα για προστασία των πεζών, κάτι που μα οδήγησε στο συμπέρασμα ότι αυτό δεν είναι ασφαλέ αποτέλεσμα. Οπότε εμεί δεν μπορούσαμε να το συγκρίνουμε με κάτι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να, κάνουμε την, για να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Δεν ξέρουμε αν λοιπόν η τραυματισμοί αυτή είναι πιο σοβαρή, παρόλο που υποπτευόμαστε ότι είναι. Ένα άλλο ερώτημα είναι ποια είναι τα μειονεκτήματα του να βρίσκεται κανεί σε ένα μικρό αυτοκίνητο αντί να βρίσκεται σε ένα μεγαλύτερο αυτοκίνητο. Ε, η απάντηση είναι ναι, υπάρχουν ε, μειονεκτήματα. Όταν κάποιο είναι σε ένα μικρό αυτοκίνητο, υπάρχουν πολλά αποδεικτικά στοιχεία που λένε ότι είναι πολύ πιο σοβαρό ο τραυματισμό. Αν δει κανεί τι μελέτε που έχουν γίνει, που είναι κυρίω από τη ΣΥΠΑ, η έκθεση και ο στόχος βεβαίως είναι πολύ διαφορετικός. 50% στις 50% ε, των ε, ε, οχημάτων είναι crossover ή μεγάλα αγροτικά οχήματα. Τώρα για την προστασία. Αυτό που κάνουμε είναι να ενθαρρύνουμε τους κατασκευαστές να κατασκευάζουν αυτοκίνητα που θα προστατεύουν το άτομο που είναι εντός του αυτοκινήτου. Αυτό σημαίνει ότι όταν σχεδιάζει κανείς το αυτοκίνητο, το, μπροστινό τμήμα του πρέπει να είναι πολύ στερεό έτσι ώστε να προστατεύεται ο, ε, ο οδηγός που βρίσκεται μέσα στο όχημα. Αν είναι τώρα το αυτοκίνητο, αυτό που γίνεται σε, ένα, σε περίπτωση ατυχήματο είναι ακριβώς και λόγω των ε, κανόνων της φυσικής όταν προκύπτει μια σύγκρουση ε, στο, στο μικρό αυτοκίνητο είναι πολύ μικρότερος ο χώρος και είναι πολύ δύσκολότερο να διαφοροποιηθεί η ταχύτητα. Και υπάρχει βεβαίως, υπάρχουν πολλά που μπορούν να γίνουν σε επίπεδο κατασκευής για να προστατευτούν οι ε, επιβάτες και γι' αυτό προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε τους κατασκευαστές προς αυτή την κατεύθυνση. Ε, άλλο ένα σημείο που ίσως να είναι λίγο απεσιόδοξο επειδή εγώ πλησιάζω τα 50. Ξέρω ότι όλοι ε, όσο μεγαλώνουμε είμαστε και πιο ε, ε, είναι και πιο πιθανό να χτυπήσουμε. Ε, οι άνθρωποι που είναι γύρω στα 52 έχουν τέσσερις περισσότερες φορές πιθανότητες να χτυπήσουν στο θώρακα από όσου είναι μικρότεροι των 52. Βεβαίως αν σκεφτεί κανείς ότι το 52 δεν είναι και τόσο μεγάλη ηλικία, ίσως είναι λίγο απεσιόδοξο το νέο αυτό. Ε, κάποια, συστάσεις τώρα, επειδή τελειώνει και ο χρόνος μου. Έχουμε μια πολύ σημαντική ε, σύσταση που θέλουμε να κάνουμε. Υπάρχουν ε, ελλείψεις στα δεδομένα για, τα, για τις συγκρούσεις και τα δυστυχήματα που έχουμε στη διάθεσή μας και καλό θα ήταν να τονιστεί αυτό και να υπάρξουν μεγαλύτερες, ε, να υπάρχουν περισσότερα ε, δεδομένα που να μπορούμε να τα συγκρίνουμε πάντως στον πλανήτη. Σε ό,τι αφορά τώρα τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν για τα οχήματα και για τους ποδηλάτες και για τους πεζούς, θα θέλαμε να ε, να δούμε ότι να υπάρχει ε, αυτόνομο σύστημα επίγουσας παίδησης στα αυτοκίνητα. Ε, υπάρχουν πολλοί πεζοί οι οποίοι δυστυχώς ε, βρίσκονται στο, στο σημείο και καλό θα ήταν να χρησιμοποιήσουμε μεθόδους οι οποίες να μπορούν να προστατεύσουν και στους δρόμους τους πεζούς. Και επίσης θέλουμε να δούμε και την ε, διεύρυνση των ε, δοκιμών που γίνονται. Όπως σας είπα πριν, ε, δοκιμάζεται κυρίως το καπότο αυτοκινήτου. Θα θέλαμε όμως να δούμε και τον 78 του 2009, τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να δούμε αν μπορεί να ενισχυθεί, να αναβαθμιστεί και να, χρησιμοποιηθεί για δοκιμές σε σημεία που όντως βλέπουμε να προκύπτουν δυστυχήματα. Πάμε τώρα στην προστασία των ε, μικρών οχημάτων. Βέβαια για όλα τα οχήματα ισχύουν, αλλά καλό θα ήταν να μιλήσουμε κυρίως και για τα μικρά αυτοκίνητα. Θα θέλαμε να υπάρχουν ε, συστήματα περιορισμού εντός των ε, αυτοκινήτων. Αυτό σημαίνει σύστημα που θα αποδίδει με τέτοιο τρόπο και θα είναι ανάλογο με, το, με, το, με τη σύγκρουση την οποία, στην οποία υπόκειται το αυτοκίνητο αυτό. Αυτό λοιπόν που θέλουμε να δούμε είναι σε μια σύγκρουση ε, όπου υπάρχει ένα ηλικιωμένο, ας πούμε ε, αυτό το σύστημα να είναι αρκετά μαλακό, ε, αρκετά ήπιο και η ζώνη ασφαλείας να είναι αρκετά ευέλικτη ώστε να μπορεί να προστατεύσει το άτομο. Αν υπάρχει πιο σοβαρή σύγκρουση, τότε ίσως να πρέπει να υπάρχει περισσότερη πίεση στην ζώνη ασφαλείας για να κρατήσει τη θέση του το άτομο. Επίσης, η, η προστασία για, τις, για το χτύπημα ε, από την πλευρά του αυτοκινήτου και τους αερόσακους. Αυτό που κάνουν οι αερόσακοι αυτοί είναι να μην ε, ε, χτυπά το κεφάλι ούτε στα πλαϊνά τζάμια ούτε στο παρμπρίζ. Και μια τελευταία σύσταση για τα οχήματα που μπορεί να δούμε συχνά στους δρόμους ε, ηλεκτρικά οχήματα τα οποία ρυθμίζονται και ε, ελέγχονται στον τύπο τους για να έχουν ε, λιγότερες προϋποθέσεις ασφαλείας. Αν όμω αρχίσουμε να, δούμε, να βλέπουμε πολύ περισσότερα τέτοια οχήματα στου δρόμου, ίσω θα πρέπει να δούμε κατά πόσο πρέπει και αυτά να υπόκεινται στου ε, κανόνε που υπόκεινται όλα τα υπόλοιπα, για να μπορούμε να έχουμε εξασφαλισμένη και την προστασία των ε, πεζών και των ε, ποδηλατών. Ε, τελευταία διαφάνεια ε, δείχνει μία έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, στην οποία συμβάλαμε και εμεί Έχει να κάνει με, τις, με τους γενικούς κανονισμούς ασφαλείας για τους πεζούς και την σκοπιμότητα τέτοιων πιθανών μέτρων. Έχουμε κάποια δεδομένα, ε, εξαιρουμένων και των δεδομένων που έχουν να κάνουν με, την, με τα πολύ βαριά ατυχήματα, που όπως σας είπα είναι λιγοστά. Ε, αν θέλετε, βεβαίω υπάρχει, μπορείτε να την έχετε στη διάθεσή σας. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κιούρντεν για την παρουσίασή σας. Δεν μπορούμε να έχουμε... Ε, τώρα, τώρα μπορούμε να έχουμε τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις, συγγνώμη. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Γνωρίζετε ότι είμαι 62 ετών, ότι κυκλοφορώ με μηχανή συχνά, οπότε είμαι πραγματικά μέρος αυτών που περιγράψατε. Πραγματικά εντυπωσιάστηκα για τους 22.000 θανάτους από αυτοκεντριστικά δυστυχήματα στην Ευρώπη. Πάντα με εξέπληκε αυτό. Τόσοι πολλοί νεκροί σε αυτοκινηστικά δυστυχήματα στην Ευρώπη. Κύριε Κέρντεν, λοιπόν, έχω τρεις ερωτήσεις για σας. Πρώτον, καταλαβαίνω αυτό που είπατε στην αρχή, ότι θα μιλήσετε για το βάρος του αυτοκινήτου. Βλέπω όμως ότι τελικά μιλάτε περισσότερο για την μορφή του οχήματος τι μορφή έχει, πώς έχει κατασκευαστεί και τι σχέση έχει αυτή η μορφή με τον πεζό. Σωστά. Έπειτα. Ταχύτητα στις πόλεις και στην Ήπεθρο. Αλλάζει. Αν έχετε αυτοκινητικό δυστύχημα στην εξοχή, με μεγαλύτερη ταχύτητα προφανώς από ότι στην πόλη που έχετε χαμηλότερη ταχύτητα. Εγώ όμω από ό,τι έχω καταλάβει, τα περισσότερα ατυχήματα γίνονται στις πόλεις. στι κατοικημένες περιοχές δηλαδή. Και τέλος, για την πόλη, τα quad που λέτε για την πόλη, τα τετράχρονα, οι τετράτροχες μοτοσυκλέτες. Μα εδώ νομίζω ότι ξεφεύγουμε. Σωστά. Όλγα Σελένοβα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Η δικιά μου ερώτηση έχει να κάνει με τις συνθήκες δοκιμής στο εργαστήριο. Σε μία από τις διαφάνειές σας αναφερθήκατε στο ότι δεν υπάρχουν αρκετά στατιστικά δεδομένα σε πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας. Το ίδιο ισχύει και για τα crash tests. Δηλαδή, διαφέρει η πραγματικότητα από τις δοκιμές στο εργαστήριο. Όπως ξέρουμε ότι συμβαίνει στην περίπτωση των δοκιμών ε, για τις εκπομπές ε, των ε, εξατμίσεων κλπ. Πώς λοιπόν μπορούμε να έχουμε σωστά στατιστικά δεδομένα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε. Η Μαρία Γκρατίνη. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη συζήτηση αυτή, γιατί είναι αλήθεια ότι η οδική ασφάλεια έχει μεγάλη σημασία για όλους μας. Ευχαριστώ πολύ επίσης και για την παρουσία σας. Ειλικρινά, περίμενα περισσότερα δεδομένα, περισσότερα στοιχεία. Τα δεδομένα που μας δώσατε είναι αρκετά γενικά, πιστεύω. Εμείς θέλουμε μελέτες με λεπτομέρειες για να ξέρουμε τελικά πώς θα νομοθετήσουμε. Με εξέπληξε επίσης που λέτε ότι τα τελευταία 15 χρόνια ο αριθμός των δυστυχημάτων μειώθηκε. Συγχρόνως όμως έχω την εντύπωση, δεν έχω βέβαια όλα τα στοιχεία, νομίζω όμως ότι ο αριθμός των ε, δυστυχημάτων, κυρίως της πόλης, αυξάνει. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας ρωτήσω, μετά από τη μελέτη αυτή έχετε να μας προτείνετε κάτι για παράδειγμα για τις επιπτώσεις των μεγάλων φορτηγών στην οδική ασφάλεια. Εγώ δεν θα μπορούσα πάντως να αποφασίσω μετά από αυτά που μας είπατε και άκουσα όσον αφορά την οδική ασφάλεια. Δεν μου φτάνουν. Ευχαριστούμε και έρχομαι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση αυτή. Η ερώτησή μου έχει να κάνει όχι τόσο με τις προτάσεις, αλλά και με κάποια άλλα πράγματα. Νομίζω ότι είναι σωστό να πούμε ότι πιο ηλικιωμένοι είναι περισσότερο ευάλωτοι από ατυχήματα. Προφανές. Γι' αυτό λοιπόν η ερώτηση μου είναι εξή: Έχουν γίνει έρευνες από όσο γνωρίζετε για το θέμα του ήχου, του θορύβου που προκαλούν τα οχήματα. Κυρίως τώρα που έχουμε όλο και περισσότερα ηλεκτρικά οχήματα στους δρόμους μας. Έπειτα, ο φωτισμός, η, τα φανάρια των αυτοκινήτων ή το χρώμα των οχημάτων επηρεάζουν καθόλου κατά πόσο δηλαδή κάποιος παρατηρεί ένα αυτοκίνητο περισσότερο από ό,τι θα παρατηρούσε κάποιο άλλο εξαιτία του χρωματός του, του φωτισμού κτλ. Έπειτα, οι νέοι κανόνες ασφάλειας σας ικανοποιούν τρόπος που γίνονται οι δοκιμές ή πιστεύετε ότι θα έπρεπε να δούμε τώρα και να βρούμε νέους τρόπους για να σχεδιάσουμε κυρίως το μπροστινό μέρος των οχημάτων. Ε, Είναι ζωτική σημασία το θέμα της οδικής ασφάλειας. Όμως στην Ευρώπη τα περισσότερα θανατηφόρα κύματα λαμβάνουν χώρα στις πόλεις μας. Σήμερα λοιπόν θα καθίσουμε να σκεφτούμε για τις πόλεις πώς θα μειώσουμε την ταχύτητα στις πόλεις. Όλο και περισσότερες πόλεις ε, δεσμεύονται για όριο ταχύτητας 30 χιλιόμετρα την ώρα. Εσείς έχετε συγκεκριμένα μέτρα, ε, συγκεκριμένα για την ταχύτητα. Αυτό είναι το πρώτο. Ο συνάδελφος μίλησε για τους ηλικιωμένους και εγώ θέλω να επανέλθω στην αυξανόμενη ούτως ή άλλως εξέλιξη που παρατηρούμε ε, μεταξύ των νέων και κυρίως των παιδιών παρατηρούμε ότι όλο και περισσότερο τα καθίσματα των αυτοκινήτων δεν είναι πλέον προσαρμοσμένα στα παιδιά. Και κοιτώντα ε, το πόσο αυξάνεται ο αριθμό των παιδιών στα ατυχήματα, υπάρχει λόγος να ανησυχούμε. Ε, επίσης να σας ρωτήσω πολύ συγκεκριμένα ε, ένας κοινός ορισμός του όρου ε, σοβαρός τραυματισμός ε, μετά από ατύχημα σήμερα δεν έχουμε τέτοιο ορισμό. Η Κομισιόν προτείνει κάποια στρατηγική για τους τραυματίες από οδικά ατυχήματα. Εσείς τι λέτε. Επίσης τι λέτε με αυτόν τον οδικό χάρτη που λέει ότι σήμερα τα κράτη-μέλη, κατάξει μιλήσαμε για τη συλλογή δεδομένων από τα σοβαρά αυτοκινητικά δυστυχήματα. Εσείς πώς θα ασκήσετε πίεση ώστε να υπάρξουν συγκεκριμένοι στόχοι μείωση του αριθμού θυμάτων σε τέτοια περιστατικά στο διάστημα 2015-2020. Ε, Συγγνώμη, μάλιστα ήρθα και αργά, δεν ξέρω αν το είπατε. Έχετε να πείτε κάτι σε σχέση με τα δικά σας στοιχεία ε, όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Οδήγησης και σε σχέση με αυτά τα θέματα. Επίσης, ε, κάνετε προβλέψεις ε, για τα αυτοκίνητα το αύριο, γιατί ξέρετε η μεγάλη πρόκληση είναι αυτό το όχημα το αύριο και το ζήτημα της ασφάλειας ε, και όχι μόνο ο ε, Για όλα αυτά τα ζητήματα λοιπόν και όλες αυτές τις φιλοδοξίες που ακούμε έχετε να μας πείτε κάτι και κάτι τελευταίο που θεωρώ αρκετά σημαντικό. Πώς προτίθεστε να υποχρεώσετε τα κράτη-μέλη να Παρατηρούν πραγματικά το ζήτημα της οδικής ασφάλειας. Παρατηρώντας τα 28 κράτη-μέλη υπάρχουν σοβαρές διαφορές. Αλλού γίνονται προσπάθειες, αλλού όχι. Ποιοι είναι λοιπόν οι δικοί σας στόχοι ώστε να ασκηθεί πίεση στα κράτη-μέλη που δεν τηρούν καθόλου τα όσα απαιτούνται από αυτά. Πώς σκοπεύετε να τους ασκήσετε πίεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είπατε ότι όσο πιο μεγάλο είναι το όχημα, τόσο μεγαλύτερο είναι και οι τραυματισμοί που περιμένουμε σε ένα δυστύχημα. Αλλά τα αυτοκίνητα γίνονται όλο πιο μικρά και πιο ελαφρά. Και 90% των δυστυχημάτων είναι ανθρώπινο λάθος. Άρα πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να αποφεύγουμε τα δυστυχήματα και να έχουμε τέτοια συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης. Αυτά νομίζω ότι μπορούν να, το, να βοηθήσουν στην κατάσταση. Έχω δίκιο ή όχι. Ευχαριστώ. Ε, Πέτερ Ευχαριστώ πολύ. Ε, καταρχάς να αναφερθώ σε κάτι που ανέφερε συνάδελφος. Είναι συγκεκριμένο το πρόβλημα όσον αφορά τα μεγάλα φορτηγά και εγώ οδηγούσα για 30 χρόνια μεγάλα φορτηγά και δεν μπορώ να πω ότι αποτελούν τόσο σοβαρό πρόβλημα γιατί ξέρετε όταν βρίσκεται κανείς ε, μέσα σε ένα μεγάλο φορτηγό δεν περνάει μέσα από αστικές περιοχές οπότε είναι λιγότερες πιθανότητες να χτυπήσει πεζούς ή ε, ποδηλάτες. Όπως είπα, έχω 30 κονταετή εμπειρία και αυτό που θυμάμαι είναι τα ζητήματα συμπεριφοράς όσον αφορά τους ποδηλάτες και τους ποδηλάτες. Του ποδηλάτες συγγνώμη και του Πεζού. Εμεί προσπαθούμε στη Σουηδία να προστατεύουμε του ποδηλάτε στο μέγιστο δυνατό βαθμό με ξεχωριστέ λωρίδε, ποδηλατόδρομου, αλλά όταν περνάει κανεί από κάποιο σταυροδρόμι, ε, συχνά η συμπεριφορά των ποδηλατών είναι απαράδεκτη. Ο κόσμο πετάγεται μέσα στη μέση του δρόμου. Και σήμερα το πρωί είδα στις Βρυξέλλες κάποιον που πετάχτηκε στον δρόμο και παραλίγο να τον πατήσει αυτοκίνητο. Ε, παρότι είχε κόκκινο φανάρι. Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα και ναι, έχουμε και το πρόβλημα των ποδηλατών. Οι ποδηλάτε πάντα θεωρούν δεδομένο ότι τα αυτοκίνητα προλαβαίνουν να σταματήσουν, αλλά αυτό δεν συμβαίνει σε όλε τι περιπτώσει. Δυστυχώ. Ξέρετε, έχουμε κάνει τόσο πολλά με τα αυτοκίνητα, τα έχουμε εξελίξει, έχουμε δημιουργήσει ε, ε, διάφορα συστήματα ασφάλειας ε, και στους δρόμους αλλά δεν ξέρω συμφωνείτε μαζί μου αυτό που χρειαζόμαστε πραγματικά είναι κάποιο είδους οδική παιδεία για τους ποδηλάτες, για τους πεζούς, για άπαντες, ώστε ο κόσμος να γνωρίζει τι μπορεί να του συμβεί εάν πεταχτεί στον δρόμο ε, όταν έχει κόκκινο ας πούμε φανάρι. Ε, πρέπει να τους εκπαιδεύσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Φυσικά είναι σημαντική συμπεριφορά και όλοι χρειαζόμαστε οδική εκπαίδευση. Ε, στην, στο Βερολίνο, ας πούμε, ε, είναι χωριστοί οι δρόμοι και είναι πολύ πιο επικίνδυνοι προφανώς ε, οι δρόμοι που είναι κοινοί όπου ε, κάποιοι ποδηλατόδρομοι τέμνονται με τους κανονικούς δρόμους και τα αυτοκίνητα χτυπούν τους, τους ποδηλάτες. Προφανώς τώρα γίνεται καλύτερη καλύτερος διαχωρισμός των δρόμων αλλά Σίγουρα δεν μπορεί κανείς να είναι ε, σίγουρος ότι κάποιος ε, οδηγός θα τον δει όσο, καλά, όσο καλή να, και να είναι η... Ε, Hat mir neulich ein, ein Vorsitzender des Autoclubs gesagt, wenn er mit dem Όσο καλός και αν είναι ο σχεδιασμός. Ένα άλλο που ήθελα να πω και είναι σημαντικό είναι η ταχύτητα. Το 30 και το 50 χιλιόμετρα την ώρα ε, στο Κοινοβούλιο προτείναμε 30 χιλιόμετρα την ώρα να μπουν στους ε, αστικούς κόμβους και μόνο όταν, ε, μπορεί κάποιος, όταν μιλούμε για δρόμους που μπορεί κανείς να τρέξει πιο πολύ να υπάρχει σαφή σήμανση. αλλά μπορεί κανείς κατά 10% να πεθάνει με το 30% και, και με 15% και με 30% συγγνώμη, ταχύτητα, με 30 χιλιόμετρα ταχύτητα να μπορεί να βρεθεί σε ένα τέτοιο δυστύχημα κατά πολύ μεγαλύτερο ποσοστό. Ε, το έχετε καθόλου εσείς ε, συγκρίνει αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, πολλές ήταν οι ερωτήσεις, θα κάνω ό,τι μπορώ για να απαντήσω σωστά. Λοιπόν, στην πρώτη ερώτηση αναφερθήκαμε στους αστικούς και στους ε, επαρχιακούς δρόμους και εκεί υπάρχει μεγάλη διαφορά. Ε, ξέρετε σε έναν ε, δρόμο υπαίθρου μπορεί να είναι πολύ υψηλότερη ταχύτητα και οι πιθανότητες επιβίωσης είναι μικρότερες. Ε, ακόμη και να επιβιώσει κανείς είναι πιθανόν να υποστεί χρόνια προβλήματα. Ωστόσο, όσον αφορά τα νούμερα, δεν βλέπουμε πολλούς πεζούς να εμπλέκονται σε ατυχήματα οδικά σε δρόμους ε, της υπαίθρου. Περισσότερο γίνεται αυτό στις αστικές οδούς. Οπότε εκεί έχουμε περισσότερα ατυχήματα σε μικρές ταχύτητες και από εκεί προέρχεται ο μεγαλύτερος αριθμός των ατυχημάτων. Τώρα η ανησυχία ότι τα έγγραφα που εξετάζουμε και οι κανονισμοί ε, ε, που αναφέρουν ε, τη σύγκρουση στα 40 χιλιόμετρα την ώρα και αφορούν την προστασία των πεζών ε, σε αυτή την ταχύτητα. Εκεί αυτές οι ταχύτητες αφορά ο σχεδιασμός. Πέραν αυτών των ταχυτήτων είναι απρόβλεπτα τα αποτελέσματα. για το άλλο ερώτημα, μιλήσαμε για τις διάφορες δοκιμές και τους κανονισμούς και με ρωτήσατε πώς αυτές οι δοκιμές σχετίζονται με τα πραγματικά περιστατικά. Σε αυτό επιμένω και εγώ διαρκώς. Χρειαζόμαστε περισσότερα πραγματικά δεδομένα. Τι έχει συμβεί λοιπόν τη δεκαετία του 70 και του 80 σε πολλές χώρες έγιναν μελέτες σε πραγματικά ατυχήματα προσπάθησαν να καταλάβουν συλλέγοντας δεδομένα τη συμπεριφορά οδηγών και ποδηλατών και πεζών ε, και αυτά οδήγησαν στους κανονισμούς που έχουμε σήμερα. Αυτό που δεν έχουμε κάνει είναι να δούμε κατά πόσο οι κανονισμοί που έχουμε θεσπίσει πραγματικά εξυπηρετούν το σκοπό για τον οποίο έχουν δημιουργηθεί. Οπότε εκεί πρέπει να εστιαστούμε στη συλλογή δεδομένων που να αντιπροσωπεύει τα περιστατικά που παρατηρούμε στην Ευρώπη. Δεν μπορώ να διαβάσω τις σημειώση μου, λέει ο μιλητή. Λοιπόν, ε, ακούσαμε μια ερώτηση όσον αφορά τη νομοθεσία και πώ μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι όλε οι χώρες θα τηρούν του κανόνε ε, συνενετικά και στα 28 κράτη-μέλη, ότι όλοι θα εφαρμόζουν του ίδιου κανόνε παντού. Ε, από την άψη των αυτοκινητοβιομηχανιών ε, αυτό είναι εύκολο διότι υπάρχει έγκριση τύπου, υπάρχουν συγκεκριμένα στάνταρ τα οποία πρέπει να τηρούνται όπω για τις εκπομπές, θέμα επίκαιρο μάλιστα. Οπότε για τα οχήματα είναι εύκολο. Αυτό που είναι πιο δύσκολο είναι η συμπεριφορά των χρηστών των δρόμων. Okay, Ακούσαμε μια σειρά ερωτήσεων για του ηλικιωμένου. Φυσικά και είναι πιο ευάλωτο, δεν σα εκπλήσει αυτό φυσικά. Αλλά αυτό που μα εκπλήσει είναι πόσο πιο ευάλωτοι γινόμαστε και πόσο πιθανότερο είναι να τραυματιστούμε σε οδικά ατυχήματα. Επίση ακούστηκε μια ερώτηση για την ηχορύπανση, τον ήχο των αυτοκινήτων λοιπόν στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που δεν υπάρχει κινητήρα σκάψη, Τι σημαίνει αυτό για του πεζού σε ένα αστικό περιβάλλον. Όταν αυτοκίνητο πηγαίνει με 40-50 χιλιόμετρα την ώρα, τα λάστιχα κάνουν περισσότερο θόρυβο από ότι ο κινητήρα. Οπότε σε αυτέ τι ταχύτητε δεν έχει σημασία αν είναι ηλεκτρικό το αυτοκίνητο ή όχι. Κάτω όμω από αυτέ τι ταχύτητε πραγματικά έχει σημασία. Οπότε πρέπει να δούμε πώ θα αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα. Πώ τα έξυπνα αυτοκίνητα θα μπορούσαν να εκπέμπουν κάποιον ήχο ώστε να προειδοποιούν τον πεζό ότι πλησιάζουν. Ε, Επίσης ακούσαμε μια ερώτηση για τα φώτα των αυτοκινήτων. Όταν ε, συζητήθηκε ο κανονισμός ε, για τους πεζούς ε, και έγινε εκτίμηση επιπτώσεων, εξετάσαμε, έγιναν δύο πράγματα. Μπήκαν στάνταρ φώτα και δημιουργήθηκε το σύστημα υποβοήθησης πέδησης, ώστε εγώ κανονικά δεν φρενάρω απότομα, ε, φρενάρω λίγο, πατάω λίγο το φρένο και το αφήνω. Έτσι συμπεριφέρεται ο περισσότερο κόσμο. στο break assist λοιπόν, το σύστημα υποβοήθηση πέδηση, ε, μεγιστοποιεί ε, τη δύναμη τη πέδηση. Έτσι λοιπόν εγκαταστήσαμε αυτό το σύστημα και τον κατάλληλο φωτισμό για τα αυτοκίνητα και πολλές μελέτες εξετάζουν το πόσο αποτελεσματικά είναι αυτά τα συστήματα. Ε, για τα ατυχήματα που σχετίζονται με μοτοσυκλετιστέ ε, κτλ. Δεν ξέρω πολλά για τι τετράτροχες μοτοσυκλέτε, δυστυχώ για τα quad, ε, οπότε δεν μπορώ να σα πω ιδιαίτερα πράγματα. Ακούσαμε μια ερώτηση. Κατά πόσο οι νέε δοκιμέ ασφαλεία που χρησιμοποιούμε σήμερα είναι κατάλληλε για τους πεζούς και για τα ποδήλατα. Παρατηρούμε ότι δεν είναι, δεν αρκούν. Έχουμε υψηλό αριθμό ατυχημάτων, ε, σοβαρών τραυματισμών σε ταχύτητες που θα μπορούσαμε να σώζουμε ανθρώπους. Ε, όταν, ε, για παράδειγμα, έχει χτυπηθεί ο πεζός από κάποιο κομμάτι του αυτοκινήτου που δεν είχε εξεταστεί στη δοκιμή. Έχουμε χρόνο ακόμα. Urban areas. Um, Για τις αστικές περιοχές ακούσαμε διάφορες ερωτήσεις για το όριο ταχύτητας στις αστικές περιοχές. 30 ε, χιλιόμετρα την ώρα είναι μάλλον ένα καλό όριο ταχύτητας. Πολλά στοιχεία αποδεικνύουν ότι στα αστικά ατυχήματα, στα, στις αστικές περιοχές όταν το όριο είναι 30 χιλιόμετρα μειώνεται ε, ο αριθμός των ατυχημάτων σε σχέση με όταν το όριο είναι 50. Φυσικά αυτό ένα τέτοιο όριο ταχύτητας δίνει περισσότερη δυνατότητα στον οδηγό να δει τον πεζό και να αντιδράσει αλλά φυσικά και η, κρούση δεν είναι τόσο, η σύγκρουση δεν είναι τόσο ισχυρή. Και μετά ακούσαμε κάποιες ερωτήσεις για τα παιδικά καθίσματα στα αυτοκίνητα. Υπάρχει ένα σχετικά νέο κανονισμός για το 1.29 για τις δοκιμές για τα παιδικά καθίσματα. Αλλά ε, είμαι ικανοποιημένο με τους κανονισμούς. Δεν είμαι πολύ ικανοποιημένο με τι κούκλε που χρησιμοποιούνται για τι δοκιμέ. Τα συστήματα συγκράτηση παιδιών ε, λειτουργούν μόνο εφόσον οι γονείς τα έχουν βάλει σωστά τα παιδιά στα συστήματα αυτά. Τα περισσότερα ατυχήματα δηλαδή, οι περισσότερε περιπτώσει ε, τραυματισμών οφείλονται στο γεγονό ότι δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά τα παιδιά στα παιδικά καθίσματα και στα συστήματα συγκράτηση. Οπότε είναι θέμα παιδεία εκεί, είναι θέμα εκπαίδευση. Επίση, ακούσαμε για το ευρωπαϊκό δίπλωμα οδήγηση. Ε, εκεί το έχασα λίγο, δεν κατάλαβα πολύ καλά, ζητώ συγγνώμη. Και μετά η ερώτηση ήταν τα ε, αυτοκίνητα του αύριο και τα αυτόνομα αυτοκίνητα, τι γνωρίζουμε για το τι θα γίνει στο μέλλον, πώς θα αλλάξουν τα αυτοκίνητα. Όσοι από εσάς έχετε παρακολουθήσει τι γίνεται με την Τέσλα, ξέρετε ε, με 2.000 ευρώ μπορείτε να επικυροποιήσετε το αυτοκίνητό σας ε, Τέσλα και να κάνει κάποιες ελιγμούς μόνο του. Υπάρχει αυτό το σύστημα το οποίο ονομάζεται αυτόματος πιλότος, autopilot. Υπάρχει διαθέσιμο φέτος Φέτος ε, αρκετοί κατασκευαστές ε, κάνουν τέτοιες δοκιμές ε, σε αυτοκίνητα στους δικούς μας δρόμους με αυτόνομα χαρακτηριστικά. Στο Λονδίνο έγινε μια έγιναν δοκιμές, θα γίνουν δοκιμές από φέτος το καλοκαίρι στην περιοχή του Greenwich. Πολλές λοιπόν μελέτες τρέχουν αυτή τη στιγμή από τους κατασκευαστές και είναι πολύ πιθανό να εμφανιστούν τα αυτόνομα αυτοκίνητα στην αγορά νωρίτερα από ό,τι περιμένουμε. Υπάρχουν κάποια νομοθετικά ρυθμιστικά εμπόδια όσον αφορά τη συνθήκη της Γενέβης, αλλά τα αυτόνομα οχήματα και η τεχνολογία αυτή από ό,τι φαίνεται είναι πιο κοντά ε, στο μέλλον από ό,τι περιμέναμε. Το τι θα συνεπάγεται αυτό για τους ανθρώπους, απουσία συγκρούσεων, διότι όπως ε, έχει διαπιστωθεί το 95% των συγκρούσεων γίνεται λόγω ανθρώπινου λάθους. Αυτό αναμένουμε, αλλά τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Ε, το 95% ε, των ανθρώπων, όπω είπαμε, ε, το 95% των συγκρούσεων οφείλεται σε ανθρώπινο λάθο και το ίδιο θα συμβαίνει και με τα αυτόνομα οχήματα. Εμεί κοιτώντα ε, συγκρούσει που γίνονταν στη Γερμανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, ε, αναπαραγάγαμε τέτοιε συγκρούσει με αυτόνομα αυτοκίνητα με αυτά τα αυτόνομα οχήματα που φρενάρουν καλύτερα. Ε, σώσαμε το 20% των ζώων, αλλά παραμένει το 80% των ατυχημάτων. Δηλαδή τα αυτόνομα αυτοκίνητα λύνουν ένα μέρο του προβλήματο, αλλά όχι όλο το πρόβλημα. Πρέπει δηλαδή να σχεδιάζουμε τα αυτοκίνητα έτσι, ακόμη και τα αυτόνομα οχήματα, με τέτοιο τρόπο, ώστε να προκαλούν λιγότερε βλάβε σε περίπτωση σύγκρουση. Μετά είχαμε μια ερώτηση για το έντα. Συμφωνώ μαζί σα. Καθώ τα αυτοκίνητα πράγματι γίνονται ελαφρύτερα, ακόμη και τα μεγάλα οχήματα ε, γίνονται πιο ελαφρά. Ε, παρατηρούμε ότι μικρύνει και το μέγεθος των αυτοκινήτων. αλλά έχουμε όλο και περισσότερα μεγάλα οχήματα στους δρόμους μας. Crossover, SUV έχουν 40% αύξηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι πωλήσει ε, τα τελευταία χρόνια. Ε, Βλέπουμε όλο και περισσότερο στο στόλο μας. Δηλαδή έχουμε όλο και μικρότερα ε, μικρά αυτοκίνητα πόλης και μεγάλα SUV και το πρόβλημα είναι σε περίπτωση σύγκρουση μεταξύ αυτών τι γίνεται. Ε, ε, τα διάφορα αυτόματα συστήματα διατήρησης λωρίδας, υποβοήθησης πέδησης, ε, εγώ υποστηρίζω πάρα πολύ αυτές τις τεχνολογίες και ε, βοηθήσαμε και εμείς την έκθεση κόστος ωφελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, σώζει πραγματικά, σώζει πραγματικά ζωές αυτές οι τεχνολογίες, τα αυτοκίνητα. Γι' αυτό θέλουμε να συμπεριληφθούν τώρα στους κανονισμούς, τουλάχιστον να συζητηθεί το θέμα αυτό. Νομίζω ότι μπέρδεψα λίγο τον κύριο από τη Σουηδία. Δεν μιλούσα για φορτηγά, μιλούσα για τα SUV, συγγνώμη. Και εσεί κάνετε κάποιε πολύ καλε παρατηρήσει όσον αφορά την εκπαίδευση, την παιδεία των ανθρώπων. Δεν υπενήσουμε ούτε κατά διάνοια ότι η εκπαίδευση δεν παίζει ρόλο. Σίγουρα παίζει ρόλο. Αλλά μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα και με τα οχήματα. Έτσι θα ήθελα να απαντήσω την ερώτησή σα. Και ε, επανέρχομαι στην ερώτηση του Προέδρου που αφορούσε την ταχύτητα και του ποδηλάτε, Και εγώ αυτό που κατάλαβα από την ερώτηση αυτή είναι κάτι στο οποίο αναφερθήκα και προηγουμένως εμείς ως άνθρωποι όταν χρησιμοποιούμε τον ε, χώρο των οδών ε, έχει σημασία η οπτική επαφή πόσο ε, είναι σημαντικό να έχει κανείς σωστή όραση να μπορεί να δει τον κόσμο και οι πεζοί να μπορούν να δουν τα αυτοκίνητα γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να ληφθεί αυτό υπόψη στη σχεδιασμό των οχημάτων Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κιούρντεν για την παρουσίασή σας, για τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις που μας δώσατε. Πάμε στο επόμενο πάνελ τώρα. Ρυθμιστικό πλαίσιο και εφαρμογή. Να δώσουμε πρώτα το λόγο στον κύριο Σάμπολ Σμιτ από τη Γενική Διεύθυνση μου. 7 λεπτά. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, ευχαριστώ πολύ που καλέσατε τις υπηρεσίες της Κομισιόν στη σημερινή ακρόαση για την οδική ασφάλεια. Θα σας κάνω μια σύντομη παρουσίαση της τρέχουσας κατάστασης και θα σας παρουσιάσω τα σχέδιά μας για το μέλλον όσον αφορά τα επιτέγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οδική ασφάλεια. Ας είμαστε σαφείς. Πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οδική ασφάλεια είναι ένας από τους τομεί όπου εκατομμύρια πολίτες καθημερινά ωφελούνται από όλα μα τα επιτεύγματα. Τα τελευταία 20 χρόνια, από τότε που ξεκίνησε η οδική ασφάλεια να αποτελεί κομμάτι του κεκτημένου, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, δεκάδε. χιλιάδε ζωέ σώθηκαν Δείτε σε αυτό το γράφημα ποια υπήρξε η πορεία τα τελευταία χρόνια και θα δείτε ότι 28.000 ζωές σώθηκαν μεταξύ του 2001 και του 2015. Όχι μόνο αυτό, είμαστε παγκόσμιοι ηγέτες σε θέματα δικής ασφάλειας, σε θέματα αριθμών. Ε, κάντε τη σύγκριση με τις ΗΠΑ. Η πιθανότητα να χάσει κανεί τη ζωή του σε ένα οδικό ατύχημα στι ΗΠΑ ε, είναι διπλάσια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, είμαστε και παγκόσμιοι πρωτοπόροι όσον αφορά τα μέσα πολιτική. Πριν δύο μήνε, τα Ηνωμένα Έθνη υιοθέτησαν στο πλαίσιο των στόχων αηφόρων αναπτύξη ένα στόχο που μοιάζει με αυτό που κάναμε εμεί πριν από 15 χρόνια όταν υιοθέτησαμε για πρώτη φορά το στόχο ε, μισών θανάτων σε οδικά ατυχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά η εξέλιξη δεν είναι ποτέ γραμμική. Έχουμε περιόδους μεγαλύτερες ή λιγότερες επιτυχίας. Αλλά κοιτώντα τα τελευταία δύο χρόνια παρατηρούμε ότι περνάμε από μια φάση επιβράδυνσης θα έλεγα και ε, στασιμότητας και αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι ότι αλλάζει το σημείο εστίασης ενώ ο συνολικός αριθμός θανάτων μειώνεται παρατηρούμε ότι το μερίδιο ευάλωτων χρηστών πεζών, ποδηλατών και μοτοσυκλετιστών το μερίδιό του το ποσοστό τους αυξάνεται. Το ίδιο και το ποσοστό των ηλικιωμένων. Αυτό βλέπουμε σαφώς. Οπότε για μας το ερώτημα είναι τώρα τι θα κάνουμε στη συνέχεια για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ε, νέες προκλήσεις και πώς θα διατηρήσουμε επιτυχή την ιστορία μας αυτή ε, δεδομένων των νέων ε, περιστάσεων. Εμείς αξιολογήσαμε την πολιτική μας, τις πολιτικές μας πέρυσι και εντοπίσαμε τρία σημεία όπου εμείς ως υπηρεσίες της Κομισιόν θα θέλαμε να συνεχίσουμε. Πρώτα απ' όλα ε, το νομοθετήματα, την νομοθετική πτυχή. Το τομέα της νομοθεσίας λοιπόν ο ε, νομοθέτης έχει κάνει ό,τι μπορούσε. Το κεκτημένο έχει ολοκληρωθεί, για να το πούμε έτσι. Μόνο ένας τομέας υπάρχει ε, που απομένει να αντιμετωπιστεί είναι το όχημα του αύριο, δηλαδή τα συνδεδεμένα οχήματα, όπου διακρίνουμε τεράστιες δυνατότητες για την οδική ασφάλεια. Γιατί αν ε, εξαλείψουμε όλο το ανθρώπινο, όλες τις πιθανότητες ανθρώπινου σφάλματος, υπάρχουν μεγάλες ε, πιθανότητες βελτίωσης της κατάστασης στο μέλλον. Είναι κάτι που μελετάμε ήδη. Πέραν αυτού εξετάζουμε και τα πιο κλασικά νομοθετήματα και εδώ αναφέρομαι στην κλασική νομοθεσία για την οδική ασφάλεια που μόλις παρουσιάσετε εσείς αλλά και τη διαχείριση της ασφάλειας της υποδομής και του επαγγελματίες οδηγούς. Θέλουμε να δούμε πού υπάρχουν αρκετά πολλές δυνατότητες βελτίωσης της νομοθεσίας ειδικότερα όσον αφορά την προστασία των ευάλωτων χρηστών των οδών που όπω είπα αποτελεί, αποτελούν όλο και μεγαλύτερο αντικείμενο ανησυχία για όλου μα. Ο δεύτερο τομέα είναι η εναρμόνιση σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν κοιτάξετε αυτό το χάρτη που έφερα για να δείτε θα δείτε μια εναρμονισμένη εικόνα. Σχεδόν όλη η Ευρώπη είναι πράσινη και πράσινο σε αυτό το χάρτη σημαίνει περίπου μέσος όρος των θανατών από αυτοκινηστικά δυστυχήματα ή και καλύτερα από το μέσο όρο. Είναι καλή εικόνα, είναι πολύ καλύτερη από ό,τι ήταν παλιότερα, αλλά από ό,τι βλέπετε υπάρχουν ε, κάποια ανησυχητικά ποσοστά ε, στα κράτη-μέλη εκείνα που έχουν μείνει πίσω σε θέματα δικής ασφάλειας. Ενώ λοιπόν λέω ότι η συνολική εικόνα είναι καλή, μπορεί να γίνει και καλύτερη. Και αυτό αποτελεί πρόκληση για όλους μας να ε, είναι πιο εναρμονισμένη η Ευρώπη. Είναι απαράδεκτο η οδική ασφάλεια να μην αποτελεί κοινή αξία ε, που επωφελεί όλους μας τους πολίτες όπου και αν ζουν. Πρόκειται λοιπόν για μια πρόκληση για όλους μας φυσικά ε, και σε εμάς την Κομισιόν. Και ξέρετε βέβαια εδώ υπάρχει, υπησέρχεται και το θέμα της επικουρικότητας. Ε, στους περισσότερους τομείς, στην εκπαίδευση, στην επιβολή του νόμου, ε, μέσω των δικαστικών συστημάτων. Εκεί έχουν αρμοδιότητα τα κράτη-μέλη. Εμείς δηλαδή μπορούμε να βοηθήσουμε μόνο περιορισμένα. Δυστυχώς δεν έχουμε ε, ειδικά κεφάλαια που να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη για την οδική ασφάλεια, αλλά βοηθούμε τα κράτη-μέλη με την ανταλλαγή εμπειριών, με συστάσεις, με την οργάνωση ειδικών ημερίδων και συναντήσεων, συνεδρίων για τα κράτη-μέλη που έχουν μείνει πίσω και φυσικά υπολογίζουμε και σε εσά ε, στους ευρωβουλευτές όταν επιστρέφετε στις ε, εκλογικές σας περιφέρειες. Αναφέρετε το ζήτημα της οδικής ασφάλειας, διότι ε, είναι μεγάλη πρόκληση ε, το να μπορέσουμε να εναρμονίσουμε όλα τα κράτη-μέλη σε ένα τομέα όπου δεν μπορούμε απλά να νομοθετούμε. Πρέπει να βασιστούμε και στη συνεργασία. Και ο τρίτος τομέας που μας αποσχολεί εμάς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το μέλλον. Ποιος είναι ο ορίζοντας πέραν της εστίασης τους θανάτους Ναι, πρέπει να λάβουμε υπόψη και τους σοβαρούς τραυματισμούς για το μέλλον. Αυτό έχει ξεκινήσει εδώ και τρία χρόνια. Ε, έχουμε αφοσιωθεί στο θέμα αυτό. Ξεκινήσαμε εξετάζοντας 17 διαφορετικούς ορισμούς του σοβαρού τραυματισμού. Τώρα έχουμε έναν ορισμό, έχουμε συγκεκριμένες μεθόδους, ξέρουμε πώς να συγκεντρώσουμε τα δεδομένα και τώρα βρισκόμαστε σε μια φάση όπου εγώ όπως κάθομαι εδώ, είμαι πολύ αισιόδοξο ότι πολύ σύντομα θα μπορέσουμε να αρχίσουμε ε, να μελετάμε τα κοινά ευρωπαϊκά στοιχεία ε, σοβαρά τραυματισμένων ανθρώπων ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα ε, τα περιστατικά αυτά διότι δεν είναι παραστατικά ήδη με αυτά των θανάτων από δικά ατυχήματα αλλά αυτή η μελέτη θα μας δώσει τη δυνατότητα να καταλάβουμε πώς προκαλούνται ε, οι τραυματισμοί αυτοί οι σοβαροί και τι πολιτική δράση χρειάζεται. Να επισημάνω και κάτι άλλο που είπαμε και στην προηγούμενη συζήτηση ότι το κύριο εντυνόμενο πρόβλημα είναι οι αστικές περιοχές, δηλαδή ακριβώς οι περιοχές αυτές όπου κανονικά λόγω της αρχής επικουρικότητας δεν μπορούμε να παρέμβουμε άμεσα. Οπότε πρέπει να βρούμε τρόπους και μέσα για να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να βελτιώσουν την οδική ασφάλεια, ακόμη και τις περιοχές εκείνες όπου εμείς δεν έχουμε άμεση αρμοδιότητα, αλλά που θα μπορούσαν ε, να γίνουν σωματικές βελτιώσεις σε θέματα οδικής ασφάλειας. Κύριε Πρόεδρε, κατάφερα να τηρήσω τα 7 λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα στην κυρία Ellen Townsend από το European Transport and Safety Council. Uh, ευχαριστώ πολύ. Εξ μέρου του Συμβουλίου για την Οδική Ασφάλεια, Σα ευχαριστώ για την πρόσκλησή μα, την πρόσκληση που μας κάνατε μας. Η οργάνωσή μα φροντίζει να δίνει ιδέε για την ε, πολιτική υπέρ της οδικής ασφάλειας. Έχω διαφάνειες, θα τις κοιτάξετε, δεν θα μπορέσω να σας μιλήσω για όλα αυτά, φοβάμαι. Λοιπόν, Θέλω να αρχίσω με κάποια νούμερα όσον αφορά τις αεροπορικές μεταφορές και τις οδικές μεταφορές. Φυσικά και θα πρέπει να μειωθούν όλοι οι θάνατοι από τις μεταφορές, αλλά να τα νούμερα από το 13 όσον αφορά τους θανάτους 25.842 και 203.500 ήταν οι θάνατοι από τα ατυχήματα αυτά, 25.000 από τα ατυχήματα. Όπως λοιπόν είπαν και οι προλαλήσαντες, δυστυχώς η κατάσταση δεν είναι καλή. Έχουμε δει κάποια επιβράδυνση βέβαια, δηλαδή έχουν μειωθεί κάπως οι θάνατοι ανάμεσα στο 2013 και το 2014, όμως χρειαζόμαστε 6,7% μείωση για να πετύχουμε την μείωση κατά το ίμιση των ε, θανάτων, των ε, θανατηφόρων ατυχημάτων, δηλαδή μέχρι το 2020. Τώρα το 2015 πετύχαμε μόνο 0,2% μείωση. Συνεπώ χρειάζεται περισσότερη δράση και σε επίπεδο χωρών μελών, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ποιε είναι οι προτεραιότητε τώρα στι δράσει μα. Η οικονομική πτυχή πρώτα απ' όλα. Γιατί πέρα από το ότι εννοείται πως ο πόνος είναι μεγάλος από τις απώλειες αυτές και το οικονομικό κόστος είναι μεγάλο. Να λοιπόν ο υπολογισμός που έχει κάνει η οργάνωσή μας η οποία εξετάζει το κόστος αν δεν είχαν σκοτωθεί όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό λοιπόν που ζητούμε εμείς είναι πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις χώρες μέλη βάσει επιστημονικών δεδομένων και βάσει συγκεκριμένων ποσοτικών στόχων. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα στην πρώτη μου δράση. Έχουμε ένα κοινό ορισμό όσον αφορά τους σοβαρούς τραυματισμούς και αυτό που ζητάει η οργάνωσή μας είναι ένας στόχος με μέτρα για την μείωση των ε, σοβαρών τραυματισμών. Η μείωση σοβαρών τραυματισμών Βέβαια δεν είναι όπως με τους θανάτους. Εδώ βλέπουμε τους υπολογισμούς που προτείνουμε, μείον 35% μείωση. Στόχος που έχει εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την ε, Λευκή Βίβλο του κ. Βατερκάμ. Επιπλέον έχουμε και νέα γραπτή δήλωση όπου μέχρι τις 18 Απριλίου και εδώ σας ζητώ όλοι να υπογράψετε πιστεύουμε ότι οι στόχοι μας μπορούν να λειτουργήσουν. Μείωση των θανάτων, αλλά μείωση και των σοβαρών τραυματισμών. Έτσι, δίνουμε νέα όθηση στις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά επιπλέον σε όλους τους τομείς που έχει αρμοδιότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση και ένας από αυτούς είναι οι προδιαγραφές των οχημάτων. Ο καθορισμός στόχου λοιπόν βελτιώνει και τον ανταγωνισμό μεταξύ των χωρών και από την μέχρι τώρα εμπειρία μας με τη συλλογή στοιχείων όσον αφορά τους θανάτους οι διαφορές μεταξύ των χωρών ε, υπάρχουν και όσο πιο πολύ επιβλέπουμε και συλλέγουμε τα αισθαστικά αυτά στοιχεία τόσο πολύ και οι χώρες σε εθνικό επίπεδο προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν καλύτερο. Η οργάνωσή μας λοιπόν έχει αυτή τη γραπτή δήλωση, συνεχίζεται η εκστρατεία μας και τις τελευταίες δέκα μέρες βλέπετε εδώ εκπροσώπους από το ETST και από το ΦΕΜΠΡ, θα ακούσετε τον συνομιλητή από το ΦΕΜΠΡ αργότερα, ήμασταν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο υψηλότερο επίπεδο με τον ε, πρόεδρο Γιούνκερ, αλλά και με τον ε, επίτροπο που είναι υπεύθυνο για τις μεταφορές. Θέλουμε ο στόχος αυτός για τη μείωση των σοβαρών τραυματισμών να προχωρήσει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή δηλαδή. Δεν πρέπει να περιμένουμε. Τώρα, να κοιτάξουμε λίγο ευρύτερα, μακροπρόθεσμα. Η Ευρώπη θέλει να φτάσει σε μηδενικά ατυχήματα. Είναι μια ιδέα που έχει έρθει από το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που εγκρίθηκε το 2011 και στη συνέχεια θετήθηκε και από την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Η οργάνωσή μας εννοείται ότι το στηρίζει. Χρειαζόμαστε διαφορετικούς ε, στόχους για διαφορετικές ομάδες και θέλουμε να υποφεληθούμε από διάφορους ε, τομείς. Έχουμε πει ότι διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν τα ατυχήματα. Να, και εσείς μερικοί κοιτάτε τα κινητά σας τώρα. Λοιπόν, υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους ο οδηγός σου μπορεί να αφαιρεθεί. Άλλη αιτία ατυχημάτων είναι υψηλή ταχύτητα, είναι το ποτό, είναι ότι δεν φοράει ε, ζώνη ασφάλειας. Πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε το θέμα της ασφάλειας στα οχήματα και την υποδομή των οχημάτων που θα ενισχύσει την ασφάλεια. έτσι ώστε να τηρούνται και οι νόμοι. Αυτοί λοιπόν είναι τομείς πάνω στους οποίους θέλουμε να δουλέψουμε. Ο τελευταίος ε, τομέας προτεραιότητας που βάζω είναι το θέμα της ασφάλειας των οχημάτων. Εσείς είσαστε ευρωβουλευτές, εκπροσωπείτε τους πολίτες, αλλά εκπροσωπείτε και τους καταναλωτές και η ασφάλεια είναι ένα θέμα κατανάλωσης. Κάθε καταναλωτής ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει εξίσου πρόσβαση σε ασφαλή οχήματα. Δυστυχώς σήμερα δεν ισχύει αυτό. Πολιούνται διάφορα οχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με επίπεδα ασφάλειας πολύ χαμηλά σε κάποιες περιπτώσεις, σε ορισμένες χώρες. Ζητούμε λοιπόν η ασφάλεια να αποτελεί μια στάνταρ προδιαγραφή. Θα έχουμε την ευκαιρία αυτή τη χρονιά με την αναθεώρηση του κανονισμού για την ασφάλεια και την προστασία να επικεντρωθούμε τα εξής θέματα που σε αυτά, ακριβώς σε αυτούς τους παράγοντες οφείλεται περισσότερη θάνατη. Λοιπόν, μείωση της ταχύτητας, κατανάλωση αλκοόλ, ο πρόσωπος από το γύρο θα σας πει περισσότερα γι' αυτό και ζώνες ασφαλείας. Τι μπορείτε λοιπόν να κάνετε Δράση σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμεί πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα συνεχή ρόλο να αντιμετωπίσει το ζήτημα. Είναι μία από τι βασικέ προτεραιότητε. Να υπάρχει λοιπόν ο στόχο για μείωση των τραυματισμών, αλλά και μετρήσει για τα αποτελέσματα των οδηγιών που ενισχύουν την ασφάλεια. Να επικεντρωθούμε στους χρήστες των κύριων αρτηριών να ασχοληθούμε με τις πιο ευάλωτες περιπτώσεις και να υποστηρίξουμε μέτρα σε εθνικό επίπεδο. Όταν μιλάτε με τους υπουργούς μεταφορών σας, λοιπόν, στις χώρες σας, πείτε τα τους όλα αυτά και βάλτε τους τα παραδείγματα, παραδείγματα από τη δικιά σας την προσωπική ζωή. Σκεφτείτε, για παράδειγμα, ότι εσείς μπορείτε να κάνετε τη διαφορά. Σας ευχαριστώ πολύ, λοιπόν, για την προσοχή σας και προσβλέπω στη συζήτηση μεταξύ μας. Ευχαριστώ την Ellen Townsend. Πάμε τώρα στον ε, κύριο Κουν Ρικούρ από την Τίσφολ. Good afternoon everybody. Καλησπέρα σε όλους και ευχαριστώ πολύ για την ε, πρόσκληση. Εγώ είμαι εδώ εκ μέρους της Τίσπολ. Η Τίσπολ είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός που ενώνει ε, όλες τις τροχές αστυνομίες της Ευρώπης. Έχουμε 28 κράτη-μέλη, ε, συν την και τη Σουηδία. Ο βασικός μας στόχος ε, είναι να σώσουμε ζωές, να αστυνομεύσουμε τους ε, δρόμους και να δημιουργήσουμε εταιρικέ σχέσεις. Από, επειδή η εικόνα συνήθως αξίζει ως χίλιες λέξεις, θα σας δείξω ποιοι είμαστε και τι κάνουμε και κυρίως τι κάνουμε για την ασφάλεια στους δρόμους.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 the slide with the human toll on our roads. Ακούσατε λοιπόν ε, για τα δυστυχήματα στους δρόμους, ε, ακούσατε και για τους εταίρους μας, για την ETSC. Συνεργαζόμαστε λοιπόν, όπως είπαμε και στο βίντεο, στενά με την Κομισιόν. Έχουμε ένα project ε, διάσωσης ζωών, έχουμε αστυνόμευση των οδών, έχουμε το project Strider, ε, για να μειώσουμε του σοβαρούς τραυματισμούς και τους θανάτου στους ευρωπαϊκούς δρόμους, κυρίως μέσω των ε, μεθόδων εφαρμογής της σχετική νομοθεσία. Επόμενη ε, διαφάνεια πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει διασυνοριακή συνεργασία, όχι μόνο διασυνορική εφαρμογή. Η διασυνοριακή συνεργασία είναι πάρα πολύ σημαντική για όλα τα μέλη. Κάνουμε 9 εβδομάδε επιχειρήσεων σε όλη τη χρονιά με, και για τα, την ασφάλεια των φορτηγών και για την ασφάλεια των λεωφορείων όπως ακούστηκε και στο βίντεο. Αν είδατε τα αποτελέσματα που έχουμε επιτύχει. Αν δείτε ας πούμε τους ελέγχους για αλκοτές, αυτές τις δύο εβδομάδες βρήκαμε, κάναμε δύο εκατομμύρια ελέγχους για αλκοτές μέσα σε δύο εβδομάδες. Μετά δεν μιλούμε μόνο για την πράξη και στην ε, θεωρία κάνουμε πολλά. Έχουμε πολλά ε, σεμινάρια, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Εδώ βλέπετε τα σεμινάρια και τις διασκέψεις που έγιναν το 2015 για την ε, ασφάλεια των δρόμων, για την τεχνολογία επίση και η μεγάλη μα διάσκεψη που γίνεται τον Οκτώβριο, που έγινε μάλλον τον Οκτώβριο, γίνεται κάθε Οκτώβριο στο Μάντσεστερ έγινε πέρσι. Η επικοινωνία είναι πάρα πολύ σημαντική για μα. Αν θέλετε να, δούμε, να δείτε περισσότερα στοιχεία για το πώ ε, εφαρμόζουμε όλη αυτή την νομοθεσία και τι κάνουμε, μπορείτε να εγγραφείτε στο ε, bulletin που στέλνουμε κάθε δύο εβδομάδες. Η προκλήση για το μέλλον, μία είναι η βασική, είναι η μείωση κατά 50% των δυστυχημάτων στου ευρωπαϊκού ε, δρόμου και προσπαθούμε να βοηθήσουμε και τον στόχο που έχει θέσει η Κομισιόν σχετικά. Αυτά, Πρόεδρε, από μένα και σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Πάμε τώρα στον επόμενο ομιλητή, τον κύριο Ζανό Μέρς από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Θυμάτων Τροχιών Ατυχημάτων. Ευχαριστώ. πολύ και ευχαριστώ πολύ που οργανώσατε αυτήν την ε, συνεδρίαση και ευχαριστώ που με καλέσατε. Συνήθως κάθομαι εκεί πίσω μπροστά από τον υπολογιστή μου, αυτή τη φορά κάθομαι εδώ. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Θυμάτων Οδικής Κυκλοφορίας κάνουμε εκστρατεία για τα δικαιώματα των θυμάτων και για την μείωση των ατυχημάτων βέβαια. Διότι θέλουμε να αποφεύγονται βέβαια οι συγκρούσεις, τα ατυχήματα, αλλά έχει μεγάλη σημασία και πώς αντιμετωπίζονται οι συγκρούσεις και τα θύματα. Αυτά τα οποία γίνονται μετά από μια σύγκρουση έχουν να κάνουν όχι μόνο με την τραυματική εμπειρία, έχουν να κάνουν και με τη δικαιοσύνη. Λοιπόν, θέλουμε να τίνουμε προς μηδενικά ατυχήματα. Το είδατε, αυτό το ακούσατε. Και θα θέλαμε να το πετύχουμε αυτό σε διεθνές επίπεδο. Είδαμε πριν με τις στατιστικές του Άλλων ότι μειώνονται οι σοβαροί τραυματισμοί και οι θάνατοι στους δρόμους. Τώρα πρέπει να επιταχύνουμε τις ε, δραστηριότητές μας και τη δράση μας. Και αυτοί που λένε ότι οι μηδενικά ατυχήματα είναι κάτι αδύνατον, θα σας πω ότι έλεγε ο Φρασίσκος της ε, Ασίζης. Έλεγε κάνε πρώτα αυτό το οποίο είναι αναγκαίο, μετά κάνε αυτό το οποίο είναι εφικτό και ξαφνικά θα καταλάβεις ότι τίποτα δεν είναι αδύνατον. Ο κύριος Σμιτ αναφέρθηκε έτσι κι αλλιώς ε, στον ΟΙΕ και στους βιώσιμους στόχους. Λοιπόν, είναι εφικτό μέχρι το 2020 να μειωθούν τα ατυχήματα κατά 50%. Θέλουμε να προσέξουμε ιδιαίτερα τους πιο ευάλωτους πολίτες, οι ηλικιωμένοι, τα άτομα αναπηρίες, τα παιδιά. Το σύστημα ασφάλειας λέει ότι όλοι κάνουν σφάλματα και ότι το ανθρώπινο σώμα, ιδιαίτερα οι πιο ευάλωτοι άνθρωποι, δεν μπορούν να αντιδράσουν έγκαιρα και να τα αντιμετωπίσουν. Γι' αυτό λοιπόν και θέλουμε να πείσουμε τους κατασκευαστές οχημάτων τα ατυχήματα να μην είναι θανατηφόρα, να προστατεύονται δηλαδή συγχρόνως οι άνθρωποι οι οποίοι μπλέκονται σε, ένα, ένα ατύχημα. Πριν από 20 χρόνια μιλούσαμε για την επιβολή κανόνων όσον αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές των οχημάτων. Τώρα μιλάμε για την ασφάλεια, δηλαδή τι υποδομή ασφάλειας μπορούν να διαθέτουν τα οχήματα σήμερα, πώς θα είναι σχεδιασμένα για τους ανθρώπους, όχι μόνο για τους οδηγούς αλλά και για τους πεζούς και για τους πιο ευάλωτους. Πρέπει να εξηγήσουμε στους πολίτες ότι δεν πρέπει να πηγαίνουν γρήγορα. Ο Άλλαν έδωσε, έδειξε ήδη κάποιες εικόνες με τον στόχο μας από σοβαρά τυχήματα. Ο Κουν δεν πρέπει να λέει απλώς να ξεπεράσουμε τα σύνορα για να μειώσουμε τους θανάτους, αλλά για να μειώσουμε και τους τραυματισμούς. Στο Λουξεμβούργο, βέβαια, έχουμε μόνο έξι ευρωβουλευτές, οπότε ερχόμαστε κάθε τρεις και λίγο και σας βλέπουμε και σας ζητάμε στήριξη, αλλά πρέπει να μας στηρίξετε και οι υπόλοιποι. Πολλά έχουν υποθεί για τα 30 χιλιόμετρα την ώρα στις πόλεις. Όντως δεν χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ταχύτητα. Βέβαια, εδώ έχουμε την αρχή της επικουρικότητας που πρέπει να σεβαστούμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως μπορεί να κάνει συστάσεις ή να παίξει ένα συμβουλευτικό ρόλο για την οδική ασφάλεια. Η Καρή Μαντάλη έφυγε τώρα, αλλά είχε τη δικιά της έκθεση για την κινητικότητα στις πόλεις, πώς αυτή θα είναι βιώσιμη. Πρέπει να συνδέσουμε λοιπόν την ε, ασφάλεια με την βιώσιμη κινητικότητα. Κάθε χρόνο 2.000 τόσα παιδιά χάνουν τη ζωή τους και 10.000 ε, τραυματίζονται. Αν ήταν τα παιδιά σας ή τα εγγόνια σας, πόσα θα δεχόσασταν να χάσουν τη ζωή τους το χρόνο. Προφανώς μηδέν. Γι' αυτό και ο στόχος μας είναι μηδέν. Θέλ, πρέπει να αλλάξουμε τις μεταφορές όχι μόνο για τα ατυχήματα, αλλά και λόγω της ρήπανση που προκαλούν τα οχήματα. Να αλλάξουμε τις μεταφορές. Σκεφτείτε ένα παιδί και έναν μεγάλο θα τους αφήνατε στον κίνδυνο, ξέρατε ότι κινδυνεύει η ζωή τους. Θα πρέπει να μειωθεί λοιπόν η κυκλοφορία στους δρόμους μας. Εδώ δεξιά βλέπετε μια ζωγραφιά από ένα σχολείο, το δημοτικό. Ένα αγοράκι ζωγράφιζε άλογα. Όντω, δεν ξέρω αν τα άλογα μπορούν να αντικατεστήσουν τα αυτοκίνητα, πάντως χρειαζόμαστε λιγότερα αυτοκίνητα. επειδή εδώ βλέπετε στην Ποκοτά ποδήλατα. Ποιο θα είναι το μέλλον τώρα των αυτοκινήτων. Τα περισσότερα έχουν περισσότερη ισχύ, περισσότερα γάλογα από όσα χρειάζονται στην πραγματικότητα και από όσα χρησιμοποιούν ιδιαίτερα στην πόλη. Γιατί να τα έχουν λοιπόν. Μαζί με άλλους ε, στηρίζουμε το Άιζα και Λάιζα που ουσιαστικά είναι ένα κίνημα που λέει ότι δεν πρέπει να εξοπλίζονται τα αυτοκίνητα με τόσο μεγάλη ισχύ εφόσον δεν τη χρειάζονται. Είναι πολύ επικίνδυνη η ταχύτητα στις πόλεις. αυτή τη γίνεται στις διαβάσεις. Λοιπόν, το Άιζα και το Λάιζα είναι ακριβώς ο στόχος μας είναι εξοπλισμός δηλαδή που εμποδίζει μεγαλύτερη ταχύτητα. Από την αρχή, από τον σχεδιασμό δηλαδή των αυτοκινήτων, τα αυτοκίνητα δεν μπορούν να αντιδράσουν επιθετικά. Αν υπήρχαν αυτά τα συστήματα λοιπόν σε όλα τα οχήματα που θα περιόριζαν την ταχύτητα, δεν χρειαζόντουσαν καν κάμερες ε, στους δρόμους που ελέγχουν την υπέρβαση ταχύτητας, όπως έχουμε και στο Λουξεμβούργο. Αριστερά βλέπετε ένα αυτοκίνητο, εντάξει δεν λέω ότι είναι για μεθαύριο, μια φωτογραφία από το Google. Πάντως εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι δεν υπάρχει καλύτερος εξοπλισμός ασφάλειας στα αυτοκίνητα από ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος. 16 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους τώρα όσοι ώρα μιλούσα, τα 7 λεπτά, και πολύ περισσότεροι βέβαια τραυματίστηκαν και ακόμα περισσότεροι υποφέρουν από τις απώλειες αυτές. Αν λοιπόν θέλετε να είστε σίγουροι ότι ηγείται στην οδική ασφάλεια η Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε θα πρέπει να βάλουμε λίγο περισσότερο πράσινο στους ε, δρόμους, αντί για το μπετόν δηλαδή και την άσφαλτο, να έχουμε πρασινάδα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για την ε, ε, παρουσίασή σας. Στην τελευταία διαφάνεια είδαμε και τον Υπουργό Μεταφορών του Λουξεμβούργου. Ακούμε τώρα την κυρία Αγιάλα Σέντερ. Eh, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δεν μπορούσα να, είμαι παρούσα εδώ από την αρχή, αλλά τουλάχιστον άκουσα τον κύριο Σμιτ και μετά. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω. Στο άμεσο μέλλον, Δεν μας μένει πια πολύς χρόνος στη θητεία μας αυτή, γι' αυτό κατεπηγόντως χρειαζόμαστε το πακέτο ασφάλειας. Και όταν ε, το λέμε αυτό, αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε την οδηγία για τις υποδομές. Επίγει. Ήδη είμαστε στο στάδιο της αυτοματοποίησης των ε, οχημάτων, του track platooning. Η υποδομή δηλαδή είναι ζωτική σημασίας. Προτείνουν η Γαλλία διάφορα τρελά σχέδια, οχήματα που θα κινούνται μόνο τους, αλλά έτσι κι ό,τι μας φαίνεται τρελό μπορεί κάλλιστα να γίνει πραγματικότητα. Τώρα οι κυρώσεις, τα πρόστιμα. Δεν προχώρησε καλά. Οπότε, γι' αυτό και χρειάστηκε συμβιβασμός από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έρθει και με το δεύτερο ήμιση, δηλαδή να είναι υποχρεωτικό να πληρώνονται τα πρόστιμα. Γιατί μέχρι τώρα είναι υποχρεωτικό, αλλά πρέπει η χώρα μέλος να ενημερώσει να φτάσει στον ε, υπεύθυνο της παράβασης, αλλά δεν έχουμε τρόπο να τον υποχρεώσουμε να πληρώνει. Ενώ χρειάζεται και αυτό. Επίσης, μας είπατε ότι δεν υπάρχει ειδικό προϋπολογισμός για την ασφάλεια. Είναι αλήθεια ότι όταν είχαμε, θα μου πείτε ότι ήταν ε, λίγα τα χρήματα, δεν τα χρησιμοποιούσαμε όμως. Ήτανε χίλιος πτέρνα. Γιατί κάθε χρόνο μας έλεγε το Ελληνικό Συνέδριο ότι δεν χρησιμοποίησαμε αυτό τον προπολογισμό. Τώρα τον έχουμε. Έχουμε το Connecting Europe Facility που μεταξύ άλλων έχει και το σκέλος της ε, ασφάλειας στους δρόμους. Θα μπορούσαμε λοιπόν να μας προτείνετε με κάποιο τρόπο να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα αυτά σε κάποιο πρόγραμμα και έτσι να μπορέσουμε να δαπανίσουμε και περισσότερα χρήματα γι' αυτό στο μέλλον. Είπατε επίσης ότι το χειρότερο σημείο είναι η πόλη. Μα ακριβώ γι' αυτό χρειαζόμαστε κι εμεί κάποιο πρόγραμμα. Ναυτιλία και πόλεις. Επίση, θέλω να ρωτήσω τον κύριο Μέρσε, έτσι δεν σα λένε, ναι. Λοιπόν, μα μιλήσατε για τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Η αλήθεια όμως είναι ότι αρχίζουμε τώρα να μπαίνουμε στην περίοδο της αυτοματοποίησης. Εγώ δεν έχω αυτοκίνητο, νοικιάζω. Όποιο αυτοκίνητο λοιπόν και αν νοικιάσω, εντάξει δεν μιλάω τώρα για τίποτα μεγάλες λιμουζίνες έτσι, έχει την... το υποβοηθούμενο παρκάρισμα, το δραβιακό τιμόνι κτλ. Άρα ο εγκέφαλος αρχίζει να δρανεί με όλους αυτούς τους μηχανισμούς. Είναι καλό. Εσείς τι πιστεύετε για αυτό τον κόσμο όπου τα αυτοκίνητα δεν ε, θα οδηγούνται από εγκεφάλους, αλλά από τον ίδιο του τον εξοπλισμό. Και σε σχέση με τρίτες χώρες πιστεύω ότι η Ευρώπη πρέπει να κάνει περισσότερο, γιατί μας το ζητάνε αυτό. Εκδημοκρατισμός, ανάπτυξη, πώς φαίνεται, από τις τουαλέτες και από την οδική ασφάλεια. Τα πεζοδρόμια, αν μπορούν οι πεζοί να κυκλοφορήσουν. Υπάρχουν χώρες που έχουν όλο και μεγαλύτερα ΑΕΠ, αλλά η οδική τους ασφάλεια είναι θανατηφόρα, θανατηφόρα για όλους, ακόμα και για αυτούς που έχουν πολύ καλά αυτοκίνητα. Το Μαρόκο μας ζητά να κάνουμε κάτι, για παράδειγμα. Έχουν δηλώσει πολύ ε, ότι θέλουν να πάρουν το λόγο, οπότε θα περιορίσουμε λιγάκι τα, τις ώρες που θα, παρα, θα παρέμβετε. Olga Silanova, Peter Lundgren und Karim Adeli auf der Liste. Äh, dann kommt als nächstes äh, Keith Taylor πρώτα. Have you worried there for a minute, Chair? Με ανησυχήσατε λιγάκι, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Δύο πολύ σύντομε ερωτήσει. Και για την ε, Κομισιόν. 30 ε, χιλιόμετρα την ώρα στις, ε, λέτε για τις αστικές περιοχές. Νομίζω ότι θα λειτουργήσει αυτό το σύστημα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση πώς μπορεί να στηρίξει την διεύρυνση αυτού του συστήματος, αυτού του ορίου. Δεύτερο ερώτημα. Αναφέρατε ότι προετοιμάζεται η αναθεώρηση του κανονισμού για την ασφάλεια των οχημάτων. Τι περιμένουμε εμείς σε ό,τι αφορά την ασφάλεια HGV, κυρίως ό,τι αφορά τους ε, πεζούς και για τους, ε, και τους ε, ποδηλάτες βέβαια. αυτά, Πρόεδρε, σύντομα από μένα. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ που ήσασταν τόσο σύντομα, Ο κύριο Έρτοκ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και όλους τους εμπειρογνώμονες στο πόντιου. Δύο ερωτήματα έχω κι εγώ. Εδώ και χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθούμε να αυξήσουμε την ασφάλεια έτσι ώστε να αποφύγουμε θανατηφόρα δυστυχήματα. Αν τώρα έγιναν οι απαραίτητες βελτιώσεις ή αν υπήρξαν, είτε πρόκειται για τους δρόμους, είτε πρόκειται για, τις, για τα αυτοκίνητα κτλ. Θα το δούμε. Ε, Βεβαίω, αν δεν εφαρμοστεί η νομοθεσία, δεν μπορεί να γίνει και τίποτα ιδιαίτερο. Οπότε σας ρωτώ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι κάνει για να ε, πιέσει τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν την νομοθεσία και δεύτερον, ε, εγώ είμαι στεναρά υπέρμαχος του να συνεχίζουμε να βελτιώνουμε τα οχήματα και από την ε, πλευρά της Κομισιόν μου λείπει ε, μια πράσινη βίβλος ας πούμε ή τέλος πάντων μια συλλογή ιδεών προς ποια κατεύθυνση πρέπει να πάμε μιλούμε για την ευθύνη, μιλούμε για την προστασία δεδομένων πρέπει πολλά πράγματα να οριστούν ακόμα οπότε καλό θα ήταν να μας πείτε αν υπάρχει κάποια τέτοια άποψη σχετικά ευχαριστώ ο κύριος Κόχα έχει το λόγο ευχαριστώ Ευχαριστώ και τους ε, παρεμβαίνοντες. Ένα ερώτημα έχω για τον εκπρόσωπο της Τίσπολ. Έχετε προβλήματα με την, ε, με, την οδηγία προστασίας δεδομένων και για την Τίσπολ αλλά και σε συνεργασία με τη Frontex, τη Europol κτλ. Ή λειτουργεί καλά η νομοθεσία και η σχετική συνεργασία. Ευχαριστώ. Τζάκι Φώστερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη που δεν ήμουν εδώ στην αρχή της συζήτησης με τον άλλο μιλητή. Έχω τρεις-τέσσερις παρατηρήσεις. Πρώτη, ε, τα ποδήλατα. Και εγώ έχω ποδήλατο και αυτοκίνητο. Και βλέπω ποδηλάτες που παραβιάζουν ε, τους νόμους, περνούν πράσινα φανάρια, δεν έχουν ε, φώτα σήμανσης και ο οδηγός τελικά του οχήματος, ε, του αυτοκινήτου ή του φορτηγού ε, βρίσκει μπελά. Πώς θα γίνει λοιπόν να δούμε τα ποδήλατα να υπάρχει κάποιο σύστημα ασφάλισης ε, για αυτά που να του το επιβάλλει αυτό. Εγώ φυσικά υποστηρίζω τα ποδήλατα. Τώρα, όσον αφορά τις αστικές περιοχές και τα ατυχήματα εκεί, έχουμε εφαρμόσει τα τελευταία 20 χρόνια ένα σωρό συστήματα από τα σαμαράκια μέχρι τις διαβάσεις και βλέπουμε ότι δεν βελτιώνεται λίγο η κατάσταση αλλά χρειάζεται και καλύτερη παιδεία στα σχολεία διότι πολύ συχνά τελικά παιδιά είναι αυτά που καταλήγουν ε, να εμπλέκονται σε τέτοια ατυχήματα. Τώρα όσον αφορά την ευαισθητοποίηση, όσον αφορά ε, την οδήγηση γενικότερα, δεν νομίζω ότι τα πρότυπα οδήγηση έχουν βελτιωθεί. Η τεχνολογία απλά έχει διευκολύνει τα πράγματα από τη δική μου άποψη. Την τελευταία 20 ετία αυξήθηκε ο αριθμό των ανθρώπων που οδηγά και δεν έχει ιδέα τι κάνει το αυτοκίνητό του και φαίνεται να οδηγούν ε, έτσι λίγο τυχαία. Θα ήθελα λοιπόν καλύτερη παιδεία, ίσως δυσκολότερες ε, εξετάσει για να πάρει κανεί το δίπλωμα. Και τέλο, θα ήθελα να πω κάτι για του αυτοκινητοδρόμου. Ναι, έχετε δίκιο η ταχύτητα, πράγματι σκοτώνει. Αλλά εγώ έχω πάει σε αυτοκινητοδρόμου με αυτοκίνητα με 30 μιλιά την ώρα στη δεξιά λωρίδα. Ε, βλέπω κόσμο να πηγαίνει εκεί και να προσπαθούν να του προσπεράσουν τα φορτηγά. Λοιπόν, το να γνωρίζει κάποιο το πώς χρησιμοποιείται ο δρόμος και να μην πηγαίνει πολύ ε, σιγά σε έναν αυτοκινητόδρομο. Ξέρετε, σε κάποιες ε, χώρες ε, έχουμε διάφορες σημάνσεις ότι βρέχει, ότι έχει σχηματιστεί ουρά. Υπάρχει τόσες πολλές σημάνσεις για τέτοια πράγματα καθημερινά και όμως που τελικά δεν ισχύουν, οπότε τελικά όταν ε, στέλνουμε ένα σοβαρό μήνυμα στον οδηγό δεν το πιστεύει. Οπότε πρέπει να δούμε πώς ε, κάνουμε όλη την επισήμανση αυτή στους αυτοκινητοδρόμους ώστε να είναι αξιόπιστη. Ευχαριστώ κύριος Κλούν. Ε, Κλούν, συγγνώμη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε πολλές πληροφορίες σήμερα, πολύ σημαντικές ε, για όλα αυτά τα ζητήματα στο πλαίσιο αυτών των προσπαθειών για οδική ασφάλεια. Χρειαζόμαστε στόχους ε, και τήρηση των στόχων. Να ρωτήσω ε, για τον τομέα των, του αλκοόλ στην οδήγηση, ποιοι είναι οι πιο αποτελεσματικοί τρόποι αντιμετώπισης του ζητήματος και των συστημάτων αυτών κλειδώματος των οχημάτων ε, Πώ ε, θα μπορούσαν να εφαρμοστούν ώστε να αποτελέσουν κομμάτι της οδική ασφάλειας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαντελή. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Με λυπεί το ότι κανένας από αυτό το πάνελ δεν αναφέρθηκε στο οικονομικό κόστος των ατυχημάτων ε, και πως αυτό επηρεάζει το κόστος της υγείας. Είναι ένα από τα πολύ σημαντικά στοιχεία για να πάμε τη συζήτηση αυτή στους αρχηγού των κρατών. Ε, Αν ναι, η Κομισιόν μου λέει δεν είναι εύκολο γιατί οι αρχηγοί των κρατών θα μου πούνε, να ξέρετε αυτό το ζήτημα, επικουρικότητα κτλ. Αλλά εσείς ω, Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχετε το ρόλο να μας πρόξετε, να μας βοηθήσετε λίγο γιατί Όλο μα λέτε, ναι, έχουμε πολλέ προσδοκίε από το Ευρωκοινοβούλιο και εγώ έχω προσδοκίε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βοηθήσει τα κράτη-μέλη και εσεί. είστε επιφορτισμένοι με τον έλεγχο σε περιπτώσει που τα κράτη-μέλη δεν εφαρμόζουν τα όσα εμείς νομοθετούμε. Οπότε για το ζήτημα αυτό τη ταχύτητα εγώ κάνω έκκληση στου συναδέλφου, επειδή είμαι για την βιώσιμη αστική κινητικότητα που αναγράφεται η ταχύτητα των 30 χιλιόμετρων την ώρα Οπότε κάντε κάτι. Έχουμε το σύμφωνο των δημάρχων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τι περιμένει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συγκεντρώστε όλου αυτού του δημάρχου και πείτε του τώρα τα πράγματα είναι σοβαρά. Μη φοβάστε, επιβάλλετε 30 χιλιόμετρα όριο ταχύτητα. Και να τελειώσω μια ερώτηση άλλη που θεωρώ ε, σημαντική. Δεν αναφέρθηκε κανεί αυτή. Κανεί δεν αναφέρεται ε, στην ευρωπαϊκή, στο ευρωπαϊκό δίπλωμα οδήγηση με νέα κριτήρια. Ε, το έχετε στα σκαριά στην Κομισιόν γιατί όταν βλέπω ότι στις διασυνοριακές συμφωνίες το λέω τώρα κατά τύχε, βλέπουμε ξαφνικά Ιταλούς ε, ε, σε ένα γαλλικό αυτοκινητόδρομο και λαμβάνουν μια, ε, ένα πρόστιμο για παράδειγμα και όσον αφορά και την ανταλλαγή ε, των στοιχείων αδειοκυκλοφορίας αυτοκινήτων μεταξύ κρατών κυκλοφορία αυτοκινήτων μεταξύ κρατών μελών, πού βρισκόμαστε ώστε να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε το ζήτημα της ε, έλλειψης ασφάλειας στους δρόμους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ε, κύριε Λούντκρεν. Ευχαριστώ θα μιλήσω αγγλικά τώρα. Μου κάνει έκπληξη που τόσος πολλοί κόσμος εξακολουθεί να μην φορά ζώνη ασφαλείας ή να οδηγά μεθυσμένος. Όλοι γνωρίζετε ότι εγώ έχω 7 αυτοκίνητα, Μ' αρέσουν πάρα πολύ, έχω και δύο αγωνιστικά. Και μ' αρέσει πολύ να πηγαίνω σε αγώνες ε, ή να οδηγώ αγωνιστικά μάλλον, τρέχοντας μέσα στο δάσος για παράδειγμα. Αλλά φυσικά ε, έχω εξοπλισμό ασφαλείας, ε, συγκεκριμένη ζώνη ασφαλείας 6 ιντσών. Αυτό είναι που θα σώσει τη ζωή σου σε περίπτωση αγώνα. Εγώ έχω πάθει πολλά σημαντικά ατυχήματα και κάθε φορά ε, βγαίνω άθικτο. Απλά λύνω τη ζώνη μου και βγαίνω από το αυτοκίνητο. Και να αναρωτιόμουν πώ γίνεται οι κατασκευαστέ αυτοκινήτων να μην έχουν αυτή την πάρα ασφαλείας ε, που έχουν τα αγωνιστικά αυτοκίνητα. Φυσικά δεν μπορεί να την έχουμε σε όλα τα αυτοκίνητα, αλλά θα μπορούσαν να έχουν μια ελαφρύτερη έκδοση ενσωματωμένη στο εσωτερικό του αυτοκινήτου αυτή τη μπάρα μπροστά, ε, προστασίας. Ε, θα μπορούσε με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσουν στην οδική ασφάλεια κατασκευαστέ. Και μετά ακούσαμε για την ίσα, ακούγεται πολύ ωραίο. Ωραίο ακούγεται, αλλά όταν ε, αναλύσει κανεί την ονομασία που σημαίνει έξυπνη προσαρμογή ταχύτητα. αυτό δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει αυτή η αντιμετώπιση μεγάλου αδερφού. Εγώ θα σας πω τι θα κάνετε. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Ευχαριστώ, κυρία Σελάνοβα. Ευχαριστώ. Το ερώτημα μου απευθύνεται στον κύριο Σμιτ και την Κομισιόν. Ε, θέλω να μου απαντήσει σε σχέση με αυτά που είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές και στο πρώτο, ο κύριος Κέρντεν δηλαδή, για την έλλειψη δεδομένων α, της πραγματικής κυκλοφορίας η Κομισιόν θα μπορούσε να βοηθήσει σχετικά. Και δεύτερο ερώτημα έχει να κάνει με το στόχο της μείωσης του αριθμού των σοβαρών τραυματισμών. Και οι τρεις ομιλητές ε, στο δεύτερο πάνελ το ανέφεραν. Και υπάρχουν και πολλοί ευρωβουλευτές μεταξύ ημών που θεωρούν ότι ο στόχος αυτός ε, για να μειωθούν ε, τα οι σοβαροί τραυματισμοί είναι πολύ σημαντικό, ακριβώ γιατί αν, δεν υπάρχει, αν υπάρχει στρατηγική και δεν υπάρχει στόχο, δεν θα είναι αποτελεσματική. Η παρουσίαση του κυρίου Σμιτ ήταν ιδιαίτερω ε, αισιόδοξη και θετική. Οπότε θα ήθελα να μας ε, πει ο ίδιος ε, ποιος είναι ο στόχος που έχει θέσει η Κομισιόν. Δεν ξέρω αν μπορούμε να δεσμεύσουμε με κάποιο τρόπο την Κομισιόν. Ε, η Κομισιόν έχει ήδη δεσμευτεί ε, να μελετήσει και τις ε, ώρες ξεκούρασης των οδηγών, να τις εξετάσει, να τις αναθεωρήσει, να τις αναθεωρήσει ίσως αναχώρα. Δεν, κανένας νόμος δεν μπορεί να εφαρμοστεί αν δεν ελέγχεται. Για την ταχύτητα επίσης το είπε και η Τζάκη Φώστερ. Φυσικά είναι σωστό να ελέγχονται και οι ποδηλάτε, γιατί όταν πηγαίνουν χωρί φω, ε, δεν καταλαβαίνω εγώ, δηλαδή πώ βγαίνουν με στη νύχτα οι ποδηλάτε χωρί ε, φω, δεν καταλαβαίνουν ότι είναι επικίνδυνο. Οι αστυνόμοι όμω δεν του ελέγχουν και στο Βερολίνο ε, δεν γίνεται κανένα έλεγχο. Έχουμε 20 αυτοκίνητα τη ε, που μπορούν να ελέγξουν την ε, την ταχύτητα και 11 λεπτά την ημέρα μπορεί το καθένα να ασχοληθεί με αυτό γιατί οι αστυνόμοι πάντα έχουν κάτι άλλο να κάνουν. Μπορεί κανείς να πάει τρέχοντας με ταχύτητα φωτός μέσα στο Βερολίνο και δεν, δεν τον ελέγχει κανείς. Αυτές είναι, αυτά είναι τα ε, αριθμητικά στοιχεία και στη Γερμανία έχουν αυξηθεί μάλιστα. Και αυτό απορρέει από το ότι δεν υπάρχει έλεγχο. Ποιε είναι λοιπόν οι δυνατότητε να παρέμβει η Κομισιόν σε τέτοιε περιπτώσει για τι για τις ώρες της επίση κάτι που θα το κάνετε, για να εξασφαλίσουμε την ε, ασφάλεια και των ε, οδηγών αλλά και των υπολείπων. Τέτοιοι έλεγχοι λοιπόν θα πρέπει να γίνονται και στι πόλει. Επειδή τώρα έχουμε πίεση για να απαντήσετε. Σας δίνουμε 2,5 λεπτά στον καθένα. Να δώσουμε πρώτα το λόγο στον κύριο Σμιτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω σε 2,5 λεπτά να απαντήσω. Για τα δεδομένα πρώτα. Θεωρώ ότι έχουμε αρκετά δεδομένα, κυρίως ό,τι αφορά τους θανάτους από τροχιά δυστυχήματα. Εκεί που έχουμε πρόβλημα είναι με την έρευνα για τα ατυχήματα, για τους λόγους που συμβαίνουν τα ατυχήματα. Εκεί αυτό είναι πάρα πολύ κοστοβόρο εγχείρημα και ευρωπαϊκά δεν έχουμε τέτοια δεδομένα. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί αυτό δυστυχώς και τα, μέτρα, και τα μέσα που έχουμε δεν είναι ε, επαρκή για να χρηματοδοτήσουν τέτοιες δραστηριότητες. Τώρα για τους σοβαρούς νομίζω ότι είμαστε όλοι στο ίδιο μήκος κύματος. Ε, η στοχοθέτηση αυτή συγκεκριμένων κατευθύνσεων έχει λειτουργήσει πολύ καλά στο παρελθόν και για τους ε, θανάτους από τα ατυχήματα θα πρέπει να δούμε πόσο στερεά είναι τα δεδομένα που μας δίνουν, πόσο αξιόπιστα είναι τα δεδομένα των κρατών μελών, τι προκύπτει από αυτά ποια είναι τα αριθμητικά στοιχεία και πότε μπορούμε να κάνουμε αυτό το βήμα ω Ευρωπαϊκή Ένωση για να θέσουμε ένα νέο στόχο. Εν τω μεταξύ όμω, τίποτα δεν μα εμποδίζει και κανεί δεν μα εμποδίζει να θέσουμε ε, ε στόχου για του ε, για σοβαρού τραυματισμού. Μπορεί το κάθε κράτο μέλο να το κάνει αυτό. Και σα ενθαρρύνω μάλιστα. Ε, να προσπαθήσω να απαντήσω και στα, επόμενα, και προηγούμενα ερωτήματα. Για τι υποδομέ για, το 30, για τα 30 χιλιόμετρα. Ε, βοηθάει ε, ώστε να αποφύγουμε τους θανάτους και τους σοβαρούς τραυματισμούς. Το ερώτημα είναι πώς θα καταλήξουμε σε αυτό και ποιος έχει την αρμοδιότητα να το κάνει. Εκεί νομίζω ότι πρέπει να θέσουμε το ερώτημα. Είναι θέμα Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό να ε, προβλέψει για κάθε κοινότητα πώς θα ρυθμίσει τα, την ταχύτητα στο ιστορικό της ή πρέπει να ενθορύνουμε την κάθε κοινότητα να πάρει σοβαρά υπόψη της αυτή την ε, νομική διάταξη και να ελέγξει, να εφαρμόσει μάλλον τη, τη ζώνη 30 χιλιόμετρων την ώρα. Και σε σχέση με αυτό, το ερώτημα της κυρία Αγιάλα Σέντερ, για να απαντήσω και όλα, είναι πολύ σχετικό. Έχουμε την οδηγία για την ασφάλεια στους δρόμους και τη διαχείριση ασφάλειας στους δρόμους και αυτή πρέπει να αναθεωρηθεί. Αν πάνε όλα καλά, στο τέλος του χρόνου, αρχές του 2017, θα είμαστε σε θέση να υποβάλουμε μια πρόταση. Αλλά αυτό είναι λίγο ακόμα, δεν είναι ακόμα σίγουρο. Ε, γιατί αυτή η οδηγία ε, περιλαμβάνει ακριβώς τέτοιες αρχές. Πριν ξεκινήσει κανείς να βάζει, να βάζει καινούριου ε, κανόνες, πρέπει να δει ποιες είναι οι συνέπειες που θα έχει αυτό που προβλέπει και νομοθετεί και πώς εφαρμόζεται αυτό στην πράξη. Ακόμα και αν αυτό εφαρμοστεί μόνο στα διευρωπαϊκά δίκτυα, αν, ε, αν το εφαρμόσουμε σωστά μια φορά και σε, έστω και σε τόσο υψηλό επίπεδο, θα μπορούσε ίσως να λειτουργήσει και σε πιο α, τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο. Επίσης, οι συνάδελφοι στη Γενική Διεύθυνση Growth δουλεύουν πάνω σε ένα μεγάλο κατάλογο διαφόρων τεχνικών προδιαγραφών, συστημάτων υποβοήθησης, ε, κυρίως για να προστατεύσουν τους ε, ευαίσθητους πολίτες. Μιλήσαμε για το όγκο, για, την, για το βάρος. Ο στόχος είναι αυτό ακριβώ να αριθμιστούν και αυτά τα στοιχεία στον κατάλογο αυτό και να υπάρξει μια πρόταση για το πώς θα πρέπει να είναι τα νέα φορτηγά και πώς μπορούμε να ε, εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των πεζών. Ε, πολλά, υπάρχουν πολλά στοιχεία που μας αναφέρατε και διάφορα συστήματα υποβοήθησης. Δεν έχουμε χρόνο να τα συζητήσουμε όμως λεπτομερώς. Το θέμα του αλκοόλ φυσικά πάρα πολύ σοβαρό θέμα η οδήγηση υπό την επίρρεια και για, το, για την εκπαίδευση για το ε, δίπλωμα οδήγηση. Ήδη από το 2000 δεν είχαμε καταφέρει να έχουμε ε, μια ε, ενιαία ευρωπαϊκή εκπαίδευση για το ευρωπαϊκό δίπλωμα, για το δίπλωμα οδήγηση. Αυτό είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Και αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να δίνουμε συστάσεις ώστε η εκπαίδευση τουλάχιστον να είναι όσο δυνατόν πιο εναρμονισμένη. Πρόεδρε, δυόμιση λεπτά μου δώσατε, καταλαβαίνετε, είναι πολύ λίγα για να απαντήσω σε αυτέ αυτές τις ερωτήσεις. Το ξέρω, παρόλα αυτά σας ευχαριστώ. Επόμενος, η κυρία Έλεν Τάουζεν. Ευχαριστώ πολύ. Για να απαντήσω στις ερωτήσεις και στα σχόλιά σας. Πρώτον, το ποτό και το δίγημα είναι ένας από τους τρεις παράγοντες που ευθύνονται για τους θανάτους στο δρόμο στα πλαίσια της αναθεώρησης της οδηγίας για την οδική ασφάλεια θέλουμε να συμπεριληφθούν όλοι οι παράγοντες. Και γιατί. Γιατί εμείς υποστηρίζουμε ότι η χρήση των, του αλκοόλ είναι τόσο επώδυνο στο τέλος πρέπει να βρεθεί ο εξοπλισμός ο κατάλληλος για να εμποδίζει τη χρήση του αλκοόλ και έχουμε διαπιστώσει ότι στις ε, περισσότερες περιπτώσεις και με τη διασυνοριακή εφαρμογή της οδηγίας δημιουργείται συνδυτοποίηση, δημιουργείται μια νοτροπία που εμποδίζει το ποτό στο δείγμα. Θέλουμε μια μεικτή προσέγγιση που να συμπεριλαμβάνει, κύριε Λούκαρντ, αυτό που λέμε εμείς μια ευφυή βοήθεια και επιμένω στο βοήθεια. Δηλαδή θα σας ενημερώνει το σύστημα για τα όρια ταχύτητας, στο δρόμο που βρίσκεστε. Και θέλουμε την αναθόρηση της ε, οδηγίας για τον εξοπλισμό ασφάλειας, γιατί πιστεύουμε ότι και έτσι μπορεί να μειωθεί η ταχύτητα στους δρόμους, όχι μόνο τους αυτοκινητοδρόμους, αλλά και στις πόλεις. Γιατί βλέπουμε ότι αυτά είναι που πρέπει να συμπεριληφθούν στη μεταρρύθμιση. Τώρα η ασφάλεια των φορτηγών. Και αυτή είναι μια προσέγγιση που θα θέλαμε να βρούμε στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φέτος και βασιζόμαστε στη δικιά σας στήριξη. Η προτεραιότητά μας λοιπόν είναι ότι οι κατασκευαστές φορτηγών θα έχουν την εντολή να σχεδιάζουν τα φορτηγά με τέτοιο τρόπο που το προστινό τους μέρος να είναι ασφαλές και για τους πεζούς που περνούν στη διάβαση για παράδειγμα αλλά και για τους επιβάτες σε περίπτωση σύγκρουσης. Όσον αφορά τώρα την εφαρμογή διασυνοριακά της οδικές, έχουμε τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κατά το παρελθόν. Περιμένουμε τώρα την έκθεση για την εφαρμογή. Ελπίζουμε να υπάρξει και συνέχεια όσον αφορά την πληρωμή των προστήμων. Συγχρόνως θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι γίνεται καλά ο έλεγχος της υπέρβασης ταχύτητας, της ε, κατανάλωσης αλκοόλ. Και περιμένουμε τώρα τα επόμενα βήματα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστούμε κύριο Σκουνδρικούρ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ακούσαμε μια ερώτηση από τον κύριο Κόχια. Αν έχουμε προβλήματα με την προστασία δεδομένων να πω ότι προκειμένου για μη κυβερνητική οργάνωση. Ε, τα, τα λειτουργικά δεδομένα περνάνε στα μέλη μας και στη Europol με την οποία έχουμε εξαιρετική συνεργασία, οπότε διευκολύνουμε τη συνεργασία και φροντίζουμε τα κράτη-μέλη να είναι ενημερωμένα. Αλλά ξέρετε για τα επιχειρησιακά δεδομένα υπάρχει και η διεθνής νομοθεσία κτλ. Τώρα για τα μέτρα έγινε μια ερώτηση για το ΆΙΖΑ. Το ΆΙΖΑ θα σήμαινε ότι θα μπορούσαμε να απαλλάξουμε ορισμένους αστυνομικού από το να ασχολούνται με την ε, τήρηση της ταχύτητας και να τους απασχολήσουμε σε άλλους τομείς ε, να ελέγχουν ε, τους χρήστε, ας πούμε κινητών τηλεφώνων που είναι ο τέταρτο παράγοντα ε, θανάτων Επίσης τώρα κανόνες καλοί μπορούν να υπάρχουν πολλοί όπως η, τα όρια ταχύτητα των 30 χιλιόμετρων στις αστικές περιοχές σε πολλά κράτη-μέλη βλέπουμε λόγω πολιτικής κρίσης ε, να μην ασχολούνται. Δεν υπάρχει επιβολή των κανόνων δικής κυκλοφορίας, ε, υποβαθμίζεται η ασφάλεια στους δρόμους. Ε, δυστυχώς ε, αυτό δεν μπορεί να γίνεται γιατί μιλάμε για το ότι σώζουμε ζωές ε, είτε ως αστυνομία είτε ως της εκπαίδευσης και η εκπαίδευση πρέπει να υπάρχει ναι θέλουμε όλοι να πηγαίνουν αργά να μην σκοτώνται κόσμο σε ατυχήματα αυτός είναι ο απότερος σκοπός Γι' αυτό λοιπόν να παροτρύνω και εσά, το Κοινοβούλιο, την Κομισιόν, να ετοιμάσετε του προπολογισμού αυτού για τα κράτη-μέλη, ώστε να ασκήσετε πίεση, ώστε η οδική ασφάλεια να παραμένει στην πολιτική ατζέντα ακόμη και σε εποχέ κρίση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Ζανό Μέρς. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα μιλήσω και εγώ γερμανικά. Υπάρχουν πολλά που μπορούμε να πούμε, αλλά σε δύο μισή λεπτά προφανώ δεν μπορούμε να τα πούμε όλα. πρέπει να προσέχουμε περισσότερο του ανθρώπου, Οι άνθρωποι κάνουν λάθη, όπω είπα και πιο πριν, σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, αλλά πρέπει να μπορούμε να διαχωρίσουμε κιόλα. για, τις, ε, για τα για τα θανατηφόρα ατυχήματα ε, είναι και το αλκοόλ, είναι και η οδήγηση υπό την υπηρεία ναρκωτικών, η έλλειψη ε, ζώνης ασφαλείας. Επίσης τα παιδικά καθίσματα είναι πολύ σημαντικά. Από το EBSR διάβασα μία μελέτη που έλεγε ότι από τα τέσσερα δεμένα με τη ζώνη παιδιά στα ε, καρεκλάκια τους, τα τρία δεν είναι σωστά δεμένα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν οι γονείς να γνωρίζουν. Εγώ ε, πάντα ε, ήμουν, φοβόμουν πολύ όταν ε, έδαινα το παιδί μου στο καρεκλάκι και προσπαθούσα πάντα να διαβάζω τις οδηγίες για να είμαι σίγουρος. Πρέπει λοιπόν να μαθαίνει κανείς από τα λάθη του να γίνει περισσότερη έρευνα για να δούμε πού γίνονται οι περισσότερες συγκρούσεις, τα ατυχήματα, πώς μπορούμε να τα αποφύγουμε για να μην τα επαναλάβουμε. Πρέπει λοιπόν να μπούμε σε βάθο. Ε, επίσης ε, πολυτομιακές έρευνες που θα μπορούσαν επίσης να γίνουν, ανταλλαγή δεδομένων, πληροφορίες, πού γίνεται τι για να μπορούμε να το αποφύγουμε την επόμενη φορά. Και επίσης ε, από την ίδια εσύ είδα μια πολύ καλή διαφάνεια με μια πυραμίδα, μια ιεραρχία. Πάνω πάνω στην, στην άκρη της, στη μύτη της ιεραρχίας βρίσκονται τα παιδιά, οι πεζοί, οι ποδηλάτες. Και αυτοί προφανώς μπορούν πολύ πιο εύκολα να τραυματιστούν Γι' αυτό πρέπει να έχουν πολύ μεγαλύτερη ευθύνη. Υπάρχουν ε, νόμοι, στην δική μου τη χώρα για παράδειγμα, πριν από δύο χρόνια ψηφίστηκε ένα νόμο, όπου ένα, αν ένα παιδί τραυματιστεί σε αστική διαδικασία, α πούμε, το παιδί προφανώ δεν έχει ευθύνη, έχει ευθύνη ο, ο, ο ενήλικα. Ίσως λοιπόν και μέσω της δικαιοσύνης δεν μπορούσαμε να λύσουμε το πρόβλημα. Επίσης για την αυτόνομη οδήγηση, θα προτιμούσα να μειώσουμε λίγο περισσότερο τη χρήση των αυτοκινήτων έτσι ώστε να μην των μηχανοκίνητων τροχημάτων για να μην καθόμαστε με τις ώρες στα, στην κυκλοφορία αλλά να κινούμαστε πολύ περισσότερο εμείς οι ίδιοι. Ε, γιατί βεβαίως πρέπει να μειωθούν τα ατυχήματα γιατί επισύρουν προφανώς και πολλά έξοδα υγειονομικής περίθαλψης μετά κτλ. Ευχαριστώ και συγγνώμη που ξεπέρασα και τον χρόνο μου. Εγώ ευχαριστώ. Πάμε στο επόμενο κομμάτι. Κατασκευαστές, ε, χρήστες δρόμου και θα ήθελα τώρα να καλέσω τους επόμενους ε, ομιλητές. Χρήστες του δρόμου, κατασκευαστές κινήτων και συστήματα υποβοήθησης ε, οδήγησης. So, um Όπως είπα λοιπόν, πάμε στους χρήστες του δρόμου, στα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης και στους κατασκευαστές. Ο πρώτος που θα πάρει το λόγο είναι ο Ματίας Κούτσεκ από την VCD. Λέσχη αυτοκινηστών στη Γερμανία. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είμαι ο Ματίας Κιούτσεκ από την VCD, Λέσχη Αυτοκινητών, στην ε, ε, Γερμανία και θέλουμε να μιλήσουμε για την βιώσιμη κινητικότητα. Και βεβαίως εμείς είμαστε υπέρ όλων ε, των ανθρώπων που είναι υπέρ της πράσινης κινητικότητας που προτιμούν να χρησιμοποιήσουν τα μέσα μας μικρής μεταφοράς, το ποδήλατό τους ή τα πόδια τους. Έχουμε κάνει πολλέ ε, εκστρατείε ασφάλειας, ε, κοστίζουν πολλά, αλλά τελικά δεν, έχουν, ε, δεν επιφέρουν πολύ, πολλά αποτελέσματα. Το ακούσαμε πολύ συχνά σήμερα και πρέπει βεβαίως να συνεχίσουμε να έχουμε ρυθμίσει μεν, τις οποίες θα εφαρμόζουμε δε. Η ασφάλεια, η ζώνη ασφάλεια εισήχθη ήδη από το, την δεκαετία του 70 και η χρήση τη. Επίσης γίνεται στην, υπάρχει στη Γερμανία πρόστιμο για την μη χρήση της ε, ζώνης ασφαλείας ε, που έχει βοηθήσει στο να φορά τελικά ζώνη ασφαλείας το 85% των ε, οδηγών και των επιβατών στο αυτοκίνητο. Ναι. Okay, nicht so Um, uh, Για το Vision Zero είναι όραμα και της Ευρώπης. Στην ε, Γερμανία όμως από το 2014 έχουν αυξηθεί ε, τα, οι αριθμοί των θανάτων και των ε, τραυματιών. Πάμε παρακάτω. Θέλουμε καλύτερη ε, ιατρική περίθαλψη. Πρέπει να υπάρξει βεβαίως ε, καλύτερη τεχνολογία για να, μιλήσουμε, για να μειώσουμε συγγνώμη, και την ε, θνησιμότητα. Πρέπει να υπάρχει καλύτερη, λοιπόν, τεχνικός, καλύτερος τεχνικός εξοπλισμός στα οχήματα. Κάτι όμως που σημαίνει ότι αυτή η τεχνολογία δίνει και μεγαλύτερη ταχύτητα στο αυτοκίνητο. Ε, αυτό λοιπόν μπορεί να, να αποτελέσει αποτελεσματικό μέτρο μόνο αν υπάρχει και ε, όριο στην ταχύτητα που ε, χρησιμοποιεί ο οδηγό, ή αν μπει ένα όριο ας πούμε στην... όταν κάνει κάποιο προσπέραση στον αυτοκινητόδρομο. Ίσως θα μπορούσαμε και εκεί να συμβάλλουμε κάπως. Θα επικεντρωθώ λίγο στη Γερμανία. Εμείς είμαστε η μόνη χώρα που δεν έχουμε όριο στην ταχύτητα στους αυτοκινητοδρόμους. Είναι ασφαλής λένε όλοι οι ε, ε, αυτοκινητόδρομοι. Ε, το μήκος τους ναι, όταν οι μετρήσεις που έχουν γίνει δείχνουν ότι είναι ασφαλής, αλλά όσο περισσότερη κυκλοφορία υπάρχει, τόσο καλύτερα είναι να υπάρχει ένα όριο τον, στην ταχύτητα. Είναι σημαντικό ο κίνδυνο. Πολύ σημαντικότερο λοιπόν ανά, ανά όχημα. πολύ πιο σημαντικό από το να μετρηθεί ο κίνδυνο αυτό ανά αυτοκινητόδρομο. φυσικά είναι καλό να υπάρχουν καλύτερε υποδομέ. Βεβαίω πάντα οι καλέ υποδομέ οδηγούν και σε υψηλότερε ταχύτητε. Οπότε η οδοπία δεν είναι στόχο θέτηση, δεν είναι στόχος αυτοσκοπός, θα πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος να ελέγχουμε την ε, ταχύτητα. Τώρα για την αποτελεσματικότητα των ε, όριων αυτών, των ορίων αυτών, συγγνώμη, έχει γίνει μια έρευνα στη Γερμανία όπου ε, μετρήθηκε ένα κομμάτι ε, του, στο Βραδεμβούργο, ένα κομμάτι του αυτοκινητοδρόμου, το οποίο παρακολουθήθηκε και ε, βρέθηκαν αρκετά σημαντικά στοιχεία. Ε, στο Βερολίνο επίσης ε, διαπιστώσαμε μια αύξηση των ατυχημάτων. Διαπιστώσαμε επίσης αυξημένη θνησιμότητα. Παρόλο που ο δρόμος ήταν καθαρός, ήταν μια μεγάλη ευθεία, για το όριο τώρα ταχύτητας, βλέπετε εδώ, το 2003 μειώθηκε και η θνησιμότητα σημαντικά το 2003, αυτά στο 0, 0 θάνατοι σε ένα χρόνο και η τάση αυτή είναι, έχει οδηγήσει σε 75% λιγότερους θανάτους και μέχρι σήμερα ε, έχουμε, αρκε... έχουμε κάπως μειούμενους αριθμούς. Ähm, ein Tempolimit in Deutschland. Το όριο ταχύτητα στην ε, Γερμανία είναι σημαντικό για δύο λόγους και για την Ευρώπη. Καταρχάς πρέπει τα οχήματα σε όλη την Ευρώπη να μπορούν να ε, να έχουν τη δυνατότητα να τρέξουν σε τέτοιες ταχύτητες για να μπορούν να, να χρησιμοποιήσουν τους γερμανικούς αυτοκινητοδρόμους, αν είναι αυτό. Και δεύτερον είναι η υψηλότερη ταχύτητα οδηγεί και σε, μεγάλη, και σε πιο δυνατές ε, μηχανές, που σημαίνει ότι ε, υπάρχει μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας εντός των πόλεων. Και αυτό σημαίνει ότι οι εκπομπές αερίων ε, διοξιδίου του άνθρακα και λοιπόν είναι πάρα πολύ υψηλότεροι και προφανώ αυτό επηρεάζει και την Ευρώπη και, τους, ε, και τη Γερμανία. Επιπλέον, Άλλο ένα σημαντικό σημείο για την οδική ασφάλεια, το είπαν πολλοί ομιλητέ, είναι αυτό το 30 χιλιόμετρα την ώρα, το όριο για τι πόλει. Είναι σημαντικό αυτό και για τον οδηγό. Ισχύει αυτό στην ε, Γερμανία. Πολλέ φορέ βεβαίω το ξεχνούμε στου ε, κύριους δρόμους. Ε, βεβαίως πρέπει να μπορεί κανεί να οδηγήσει μέχρι 50 ε, χιλιόμετρα, αλλά αν δεν, υπάρχουν, ε, αν δεν υπάρχει σήμανση, πρέπει ο οδηγό να ξέρει ότι επιτρέπεται μέχρι 30. Αυτό πρέπει να είναι το όριό του και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, Σημαντικό είναι να σκεφτούμε ότι 95% των ατυχημάτων γίνονται με, προκαλούνται από τον οδηγό και εμπλέκουν πεζούς ή παιδιά. Υπάρχει μια μείωση, υπάρχει δυνατότητα να, μειωθούν, να μειωθεί αυτό το ποσοστό και θα πρέπει κανείς να σκεφτεί και ότι δεν υπάρχει άλλο όχημα το οποίο να, ε, δεν εγκρίνεται κανένα άλλο όχημα ή καμία άλλη συσκευή που να προκαλεί 22.000 θανάτους το χρόνο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να το έχουμε στα υπόψη μας για την οδηγή, την ασφάλεια. Εμείς λοιπόν προτείνουμε να υπάρχει ένα όριο ευρωπαϊκό 130 ε, στους ε, αυτοκινητοδρόμους, 30 στις πόλεις για να προστατεύσουμε και το περιβάλλον και επίσης ε, πρέπει να υπάρξει μετάβαση στους σιδηροδρόμους από, τους, από τα φορτηγά, ε, ειδικά από τα βαρέα φορτηγά, ε, αυτά που είναι πάνω από 1,5 τόνο. Ίσως αυτά να πρέπει να έχουν δικό τους όριο ταχύτητας. Για τα λιγότερο βαριά ε, φορτηγά επίσης πρέπει να υπάρξει μια μετάβαση προς τους σιδηροδρόμους και επίσης πρέπει να υπάρξουν πάρα πολύ αυστηρά όρια στο αλκοόλ και στους ελέγχους που γίνονται για το στο, με το αλκοτέστ. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής ο κύριος Παύλο Νούνες Δεμούρα από την Γιροκέρ. Να σας ζητήσω να αλλάξετε τις διαφάνειες. Καλησπέρα σε όλους. Το όνομα μου είναι Παλό Νούνες Δεμουρά και είμαι υπεύθυνος πολιτικής στην Eurocare που έχει έδρα τη Βρυξέλλης. Εδώ βλέπετε την ιστοσελίδα της Eurocare. Είμαστε μια συμμαχία με κυβερνητικών οργανισμών δημοσίας υγείας για την πρόληψη και τη μείωση των βλαβών που προκαλούνται από, από το ενόπνευμα στην Ευρώπη. Έχουμε 60 οργανισμούς μέλη από 30 ευρωπαϊκές χώρες. Το ζήτημα του αλκοόλ είναι ευρύ. Επίσης ασχολούμαστε ε, συγκεκριμένα με την οδική ασφάλεια. Όπως βλέπετε στην κορυφή της σελίδας ε, υποστηρίζουμε το έργο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την οδική ασφάλεια και επίσης υποστηρίζουμε και το έργο των ε, συναδέλφων της ETSC του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ε, Ασφάλειας Μεταφορών. Πιο συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή ε, υποστηρίζουμε, υποστηρίζουμε την εκστρατεία του ETSC καθώς αυτό κάνει έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει έναν ε, πολύ αναμενόμενο στόχο μείωσης των σοβαρών τραυματισμών στους δρόμους. Έχουμε συγκεκριμένες ε, ε, προτάσεις και συστάσεις πολιτικής για την οδήγηση υπό την επίρρεια. Εδώ βλέπετε μια σύνοψη, ουσιαστικά μηδενική ανοχή Πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει ασφαλής ποσότητα αλκοόλ. Όταν οδηγεί κανείς δεν πρέπει να πίνει σε καμία περίπτωση, καθόλου. Επίσης θέλουμε μεγαλύτερη εναρμόνιση. εναρμονισμένα όρια, ανώτα όρια σε ολόκληρη την Ευρώπη. Επίσης, ε, μας απασχολεί το ζήτημα της επιβολής των νόμων. Θεωρούμε ότι εφόσον υπάρχουν νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται και πρέπει να ε, αφιερώνονται σε αυτό συγκεκριμένοι πόροι. Και για όλα τα αλκοτέστ επίσης. Ε, χρειαζόμαστε επίσης ένα αρμονισμένο σύστημα ε, ποινών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Επίσης προτείνουμε ενημέρωση κατά τα μαθήματα οδήγησης, ε, τις εξετάσεις οδήγησης ε, και οι πληροφορίες αυτές να δημοσιεύονται σε όλες τις ε, σχολές οδήγησης. Θέλουμε απαγόρευση πώληση υνοπνευματοδών σε πρακτήρια βενζίνης και σε καταστήματα αυτοκινητοδρόμων. Επίσης ε, θέλουμε να υπάρχουν συστήματα κλειδώματο και κινητοποίηση των οχημάτων ε, με μέτρηση της αλκοολεμία ε, για τους επαγγελματίε οδηγού, και όσους έχουν ήδη βρεθεί να οδηγούν υπό την επίρρεια Επίσης θέλουμε επισήμανση και στις ε, συσκευασίες των υλοπνευματοδών. Θέλουμε δηλαδή ο τομέας των υλοπνευματοδών να ενημερώνει τους καταναλωτές για τους κινδύνους της οδήγησης υπό την επίρρεια. Προηγουμένως αναφέρθηκα ε, στις συγκεκριμένες ε, συστάσεις που έχουμε σε ακριβές συστάσεις μείωση των βλαβών από το αλκοόλ στον τομέα της οδήγησης υπό την επίρρεια. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και τις ευρύτερες συστάσεις. Όσον αφορά την οδήγηση υπό την επίρρεια, οι προτεραιότητες φαίνεται να είναι η διαθεσιμότητα και η επιβολή του νόμου και φυσικά η ενημέρωση. Αλλά ξέρετε έχουμε ένα πρόβλημα με την ε, βιομηχανία ενοπνευματοδών. Όλοι μας ε, όπως ξέρετε εδώ υποστηρίζουμε ότι δεν πρέπει κανείς να πίνει κανονικά. Ε, η βιομηχανία μας των πνευματοδών υποστηρίζει εμάς τις προσπάθειές μας αυτές, μείωση της χρήσης αλκοόλ κατά την οδήγηση, αλλά ταυτόχρονα υποσκάπτει τις προσπάθειες αυτές. Τις ευρύτερε προσπάθειες που θα έπρεπε να καταβάλουμε για να μειώσουμε τις βλάβες από το αλκοόλ, για παράδειγμα. Ο Παγκοσμίος Οργανισμός Υγείας επίσης και όσα λένε ότι ε, η τιμή ε, παίζει σημαντικό ρόλο και η βιομηχανία των πνευματοδών. Ε, ξέρετε, αυτά είναι δύο παραδείγματα. Τσακώνται τώρα με τις, με τις σκοτσέζικες αρχές και θέλουν να εισάγουν συγκεκριμένες τιμές βάσει συστάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας. Και η βιομηχανία των ενοπνευματοδών προσπαθεί να βάλει εμπόδια ε, σε αυτή την εισαγωγή τιμής μονάδας ε, ε, στη Σκωτία όπως είπα. Ένα άλλο παράδειγμα που δεν έχει ακόμα σχέση με την νομοθεσία αλλά πρόκειται για ένα πρόβλημα ως εξή. Είναι ένα πρόβλημα αν μη τι άλλο ηθικής. Η βιομηχανία των υνοπνευματοδών και εδώ αναφέρομαι μόνο στα πιο βαριά είναι προβληματόδη είναι χορηγοί της Φόρμουλα 1 και έτσι δημιουργούν ε, μία, ένα συσχετισμό μεταξύ του αλκοόλ και της οδήγησης αλλά όχι μόνο και της οδήγησης αλλά και της υψηλής ταχύτητας πιστεύουμε ότι αυτός ο συσχετισμός ε, δεν θα έπρεπε να λαμβάνει χώρα Θέλουμε λοιπόν να αποσυρθούν από τις χορηγίες αθλητικών αγώνων αυτοκινητιστικό και ειδικότερα της Φόρμουλα 1. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Gian Franco. The Mobile Manufacturers Association. Μπούτσιο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα κυρίε και κύριοι. Και σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να συμμετάσχω στη συζήτηση αυτή εκ μέρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων. Εδώ βλέπετε τα μέλη μας. Μια εταιρείε εμπορικών αυτοκινήτων. Στο διάγραμμα αυτό βλέπετε ποια είναι η γενική τάση όσον αφορά τα ατυχήματα, τους τραυματισμούς και τους θανάτους. Είναι θετική η τάση, όπως έδειξαν και οι συνάδελφοι πριν από μένα. Πρέπει όμως να κάνουμε περισσότερα. Εδώ κοιτάμε τον αριθμό των θανάτων σε σχέση με τα χιλιόμετρα που διανύουν το χήματα. Βλέπετε λοιπόν ότι στην Ευρώπη κατά μέσο όρο έχουμε 59 ε, θανάτους για 10 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Βέβαια η διαφορά είναι τεράστια από χώρα σε χώρα. Στη Σουηδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο τα πράγματα είναι καλύτερα συγκριτικά με άλλες χώρες από τις ίδιες συνθήκες δηλαδή όσον αφορά τον αριθμό των οχημάτων που κυκλοφορούν, τις υποδομές, τους δρόμους κτλ. Όπως για παράδειγμα είναι η Αυστρία και το Βέλγιο. Τρία στοιχεία μπορούν να συνεισφέρουν στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Ο οδηγός, η υποδομή των δρόμων και το όχημα. Χρειάζονται λοιπόν στρατηγικές για να αντιμετωπιστούν και τα τρία αυτά στοιχεία. Εμείς πιστεύουμε ότι όπως δείχνουν και τα στοιχεία που σας έδειξα, τα ωφέλη από μη τεχνικές λύσεις, υποδομές δηλαδή οχήματα, δεν έχουν τύχη επακούς εκμετάλλευσης. Για παράδειγμα, στην, στις διαφάνειες αυτές βλέπουμε στη Σουηδία την εισαγωγή κάποιων τεχνητών διαχωριστικών σε δρόμους της Υπέθρου να αποτέλεσμα να τιμήσει κατά 60% τον αριθμό των θανάτων. Υπάρχουν όμως και λύσεις που ονομάζουμε ενεργούς ασφάλειας. Τι σημαίνει. Σημαίνει ε, ότι μπορούμε να έχουμε συστήματα ε, αυτόματης πέδησης του οχήματος ή ειδοποίηση σε περίπτωση αλλαγή λωρίδας κτλ. Αν επεκταθούν αυτά τα συστήματα μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση και εμείς προτείνουμε να συζητηθούν στα πλαίσια της αναθεώρησης της οδηγίας. Πρέπει βέβαια να υπάρχει και ρεαλιστική δοκιμή των συστημάτων αυτών. Σήμερα υπάρχει η τεχνολογία για να βοηθηθεί ο οδηγός να ενημερωθεί για την ταχύτητά του, για την υπέρβαση ταχύτητας. Πρέπει όμως να έχουμε ομοιόμορφα κριτήρια όταν ορίζουμε όρια ταχύτητας και η υποδομή του δρόμου πρέπει να είναι αντίστοιχη ώστε να μπορεί να περνάει η ενημέρωση στον οδηγό ανάλογα με την υποδομή του δρόμου. Τώρα, το ποτό και οδήγηση βέβαια είναι κάτι πολύ σοβαρό. Υπάρχει σήμερα κατάλληλη τεχνολογία για να αποφύγουμε να αρχίσει να μπει στο αυτοκίνητό του και να ξεκινήσει ένας οδηγός εφόσον έχει υπερβεί κάποια επίπεδα αλκοόλ στο αίμα του. Γίνεται, υπάρχει τέτοια ειδοποίηση, αλλά ακόμα δεν είναι αποτελεσματικό και δεν είναι κάτι απόλυτα αποδεκτό από τους οδηγούς. Δεν το θέλουν όσοι δεν κάνουν κατάχρηση αλκοόλ, που είναι και περισσότεροι. Ε, βρέχει πρόθεσμα πάντως, μπορούν τα οχήματα να εξοπλιστούν με ένα σύστημα το οποίο κλειδώνει το αυτοκίνητο σε περίπτωση κατανάλωτης αλκοόλ. Υπάρχουν και άλλες πιο μακροπρόθεσμες ε, λύσεις και εδώ βλέπετε τον κατάλογο των εταιριών που συμμετέχουν σε τέτοια προγράμματα για να αναπτυχθεί η τεχνολογία εκείνη η οποία θα βοηθήσει χωρίς καθυστέρηση να υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός χωρίς να πρέπει ο οδηγός να κάνει τίποτα ιδιαίτερο. Τέλος, πριν καταλήξω, η τελευταία μου διαφάνεια αυτή δείχνει ποια είναι η τάση όσον αφορά το μέσο όρο ηλικία των οχημάτων που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 10 ετών είναι σήμερα. Βέβαια, όταν η τεχνολογία είναι στάνταρ, θα χρειαστούμε 10 χρόνια ώστε να έχουμε 50% των οχημάτων ξεπλυσμένων με τη... τα αισθήματα δικής ασφάλειας. Συμπεράσματα. Πρώτον, βελτιώσεις μπορούν να υπάρξουν και ωφέλη για την ε, οδική ασφάλεια αν αλλάξει η συμπεριφορά και οι υποδομές. Δεύτερον, η παθητική ασφάλεια μπορεί να βελτιωθεί και να αντικαταστεί σιγά σιγά με την ενεργό ασφάλεια. Έπειτα, οι υποδομές μπορούν να βελτιωθούν. Έπειτα, η συμπεριφορά του οδηγού που τότε έχουμε άμεσα ωφέλη. Ενώ για την υποδομή, όπως είπαμε, χρειάζονται 10 χρόνια για να έχουμε 50% βελτίωση. Έπειτα, τα οχήματα κατασκευάζονται έτσι που να μπορεί να υπάρχει συνεργασία. Έπειτα, ο αυτοματισμός, όπως είπαν και οι συνάδελφοι πριν, μπορεί να προσφέρει τεράστια ωφέλη μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα στην οδική ασφάλεια. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Εγώ ευχαριστώ. Ε, τελευταίος ομιλητής, ο Σεμπάστιαν Φέλτμαν από τη Ρόλαντ Μπέργκερ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Θέλω λίγο να σα επιστήσω την προσοχή στα, στις ε, πτυχές της τεχνικής και της ρύθμισης ό,τι αφορά την υποβοήθηση και την αυτόνομη οδήγηση. Αρχικά να πω δύο σύντομα λόγια για τη Roland Berger από το, ιδρυθήκαμε το 68, ε, είμαστε συμβουλευτική εταιρεία ε, για πολλές άλλες εταιρείες. Ε, προσπαθούμε να έχουμε ανεξάρτητες γνωμοδοτήσεις για τα θέματα κινητοκότητας, υποβο, υποβοήθησης οδήγησης, αυτόνομης οδήγησης. Κάτι που θεωρούμε ότι μπορούμε, μπορεί να εφαρμοστεί και σε ευρωπαϊκή πλήμμα και θα ήθελα να σας πω δύο πράγματα σχετικά κάποια αρχικά αριθμητικά στοιχεία. Είναι πραγματικά τρομακτικά τα νούμερα, το πώς θάνατοι υπάρχουν στην Ευρώπη. Σε πόσες περιπτώσεις τώρα ένα άτομο είναι αυτό που προκαλεί το ατύχημα. Οι τα τελευταία δεδομένα λένε ότι 90% όλων των ατυχημάτων είναι, έχουν αιτία το ανθρώπινο λάθος. 76% είναι ε, το άτομο το ίδιο αυτόματο, ε, υπεύθυνο για αυτό που έχει συμβεί. Μιλήσαμε για, ε, για την κούραση, για την έλλειψη προσοχής, ε, για την απειρία, επίσης το, το αλκοόλ και το τιμόνι. Είναι πολλοί οι παράγοντες που οδηγούν τελικά στο να ε, μην μπορεί κανείς να οδηγήσει, αλλά να μην μπορεί και να φερθεί έξυπνα, έστω και αν βρίσκεται επί την επίρρεια όλων αυτών. Η ψηλή ταχύτητα επίσης είναι σημαντικός παράγοντας. Η τεχνολογία βεβαίως ε, πολλές φορές ε, βοηθάει, ε, η τεχνολογία προχωράει και έχουμε δει σε ποιους τομείς μπορεί κανείς να μιλήσει για αυτόνομο για αυτόνομη οδήγηση. Η αυτόνομη οδήγηση είναι σίγουρα κάτι που θα υπάρξει σίγουρα και στο μέλλον. Βεβαίως είναι ένας από τους παράγοντες που επηρεάζει τα πράγματα. Έχουμε κάνει μια έρευνα για το θέμα της αυτόνομης οδήγησης, της αυτόματης οδήγησης, διαπιστώνουμε σήμερα ότι υπάρχουν ε, πολλά κλασικά είδη κινητικότητας ε, από ταξί ή άλλα οχήματα που προκαλούν ε, ατυχήματα. Υπάρχει μια μεγάλη αγορά που βρίσκεται μπροστά μας ε, από χώρες, από οργανώσεις, από επιχειρήσεις ε, που βάζουν ε, δισεκατομμύρια. Μάλιστα πρόσφατα το 2017 μας είπαν, μας είπανε κάποιες αυτοκινητοβιομηχανίες στη Γερμανία ότι θα επενδύσουν 3 δις ευρώ για να προωθήσουν την αυτόματη οδήγηση. Τώρα, αν μιλήσουμε για την Ευρώπη και, τη, και τα συστήματα υποβοήθησης, οι κατασκευαστές έχουν αποφασίσει να έχουν ε, πλήρη ε, εισαγωγή του συστήματος αυτού, βεβαίως έχοντας υπόψη και την ασφάλεια των, ε, της οδήγησης. Πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ από Ευρωπαίους κατασκευαστές επενδύθηκαν στην, στα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό ποσό και αν δούμε το δίκτυο για, τον, για την αυτόματη οδήγηση που βλέπουμε ανά τρίμηνο, οι, οι Γερμανοί, οι, γενικώ οι Ευρωπαίοι ας πούμε, ε, κατασκευαστές, το θέμα της τεχνολογίας για την υποβοήθηση και την αυτόματη οδήγηση είναι πραγματικά πολύ σημαντικό για αυτούς και βεβαίως χρειάζεται την δική σας στήριξη. Είχα πει ότι θα σας, κάνω, θα σας δείξω έναν μικρό οδικό χάρτη για το τι γίνεται η οδήγηση και πώς θα εξελιχθεί. Να σας θυμίσω ότι μιλούμε για ε, το ερώτημα πώς ε, μπορούμε να αποφύγουμε την, ε, τέτοιου είδους ε, προβλήματα, πώς, μπορεί δηλαδή να, πώς μπορούμε να προκαλέσουμε την ενεργό ανταπόκριση του οδηγού. Στο δεύτερο μιλούμε για το τι γίνεται με, την, ε, με κάποια πούμε βαρετή κατάσταση που μπορεί να βρεθεί ένας οδηγός στον αυτοκινητόδρομο ή να μην έχει την προσοχή του εστιασμένη και να προκαλέσει ατύχημα. Τι γίνεται με τις υποδομές επίσης των αυτοκινητοδρόμων, πάρα πολύ σημαντικό θέμα και προκύπτει σε πολλές ε, ε, συζητήσεις και σε πάρα πολλές επίσης ε, ξεχνιέται. Και ένα ε, σχόλιο εδώ. Αν μιλούμε για την ε, επικοινωνία car to car, το αυτοκίνητο, το όχημα γίνεται ένας παίκτη της ομάδας ουσιαστικά. Α πούμε μπορεί να, έχει, να έχουν υπάρξει προειδοποίησει για πάγο ή για χιόνι ή για κρύο. Αυτό θα μπορεί μέσω τη τεχνολογία ίσω να οδηγήσει και σε μείωση τη ταχύτητα. Είχαμε πολλές περιπτώσει όπου βρίσκονται πολλές ε, προειδοποιήσεις ε, για πάγο ή για χιόνι, σε πολλά αυτοκίνητα ήδη υπάρχουν ε, τέτοιες, ε, τέτοιες δυνατότητες. Μπορεί κανείς ε, πλέον να παρκάρει και το αυτοκίνητό του χωρίς να χρειάζεται καν να είναι μέσα στο αυτοκίνητο και πίσω από το τιμόνι. Το αυτοκίνητο, το τιμόνι λειτουργεί από μόνο του και παρκάρει το αυτοκίνητο. Υπάρχουν πολλέ λοιπόν καινοτομίε ε, από την πλευρά τη τεχνολογία ε, και είναι διαθέσιμε, οι οποίε βεβαίω ε, πρέπει να υπόκεινται σε κάποιε ρυθμίσει, τουλάχιστον στον ευρωπαϊκό χώρο. Μιλούμε για την πλήρω ανεξάρτητη, αυτόνομη συγγνώμη, οδήγηση για μια περίοδο από το 2020-2025, πιο πριν δεν μπορεί δηλαδή να γίνει κάτι τέτοιο. Κλείνοντας να πω, εσείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πώς μπορείτε να βοηθήσετε σε ό,τι αφορά την ε, εισαγωγή των αυτόματων αυτών συστημάτων. Καταρχά, η διασύνδεση είναι πάρα πολύ σημαντική και βεβαίω πρέπει να ενισχύσουμε την ασφάλεια στους δρόμους. Φυσικά υπάρχει θέμα εδώ πολιτική παρέμβαση, πολιτική βούλεση για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε το πλήρε φάσμα της τεχνολογίας. Πρέπει βεβαίω να είμαστε ε, ενήμεροι για τι τεχνικέ ε, εξελίξει και οι καινοτομίε βεβαίω δεν πρέπει να αποτρέπονται. Πρέπει να υπάρχει μια ασφάλεια δικαίωση σε όλη την Ευρώπη. Βεβαίω ε, αυτό πρέπει να γίνει συνολικά. Ε, αυτά είναι κάποια από τα θέματα τα οποία εμένα με ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Η πιστοποίηση των οχημάτων, ε, τι γίνεται ας πούμε με το Audi και γιατί μπορεί να κυκλοφορήσει με πολύ περισσότερες ε, με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα την ΣΥΠΑ αντί για την Ευρώπη, γιατί στη ΣΥΠΑ υπάρχουν πολύ περισσότερες δυνατότητες για δοκιμές ε, για τέτοια συστήματα υποβοήθησης οδήγησης. Ε, δεύτερον, ρύθμιση, το είπα ήδη. Ε, κατά την άποψή μας ε, είναι καταστροφικό ότι ακυρώθηκε η σχετική συμφωνία και δεν αναπληρώθηκε από κάτι. Είναι ε, παροχημένη η ε, συμφωνία αυτή βέβαια και πρέπει να ανανοηθεί ασφάλεια και αποφυγή ατυχημάτων. Όλοι συμφωνούμε ότι ποτέ δεν μπορούμε να έχουμε 100% ασφάλεια όσο και αν ε, ένας άνθρωπος οδηγεί ή οδηγεί το αυτοκίνητο με το αυτόματο σύστημα ή ό,τι και γίνει δεν μπορούμε να έχουμε 100% ασφάλεια αλλά αντί να μιλούμε για ηθικές προσεγγίσεις και να κάνουμε φιλολογικές συζητήσεις και όλο θα ήταν να δούμε ότι πρέπει να υπάρχει ένας ρυθμισμένος χώρος, ένα πλαίσιο ασφάλειας, όπως υπάρχει το, η Αμερικανική Αρχή Οδικής Ασφάλειας, που βάζει μαύρα κουτιά στα οχήματα. Εμείς συμφωνούμε με αυτό όπως έχουν τα αεροπλάνα. Ίσως έτσι να δούμε ε, κατά πόσο υπάρχει πρόκληση ατυχήματο ε, από ε, εξωτερικούς παράγοντες. Τέταρτο σημείο, δεδομένα και προσωπικά δεδομένα. Προστασία των δεδομένων και έχουν συμφωνήσει για κάποιες αρχές ό,τι αφορά τη διαφάνεια, την διάθεση και την ασφάλεια των δεδομένων. Η συζήτηση νομίζω ότι έχει διεξαχθεί πολύ επικοδομητικά. Βεβαίω πάντα υπάρχει το θέμα του νομικού πλαισίου το οποίο παραμένει εκρεμέ. Ευρωπαϊκά ε, θα πρέπει και οι κατασκευαστέ ε, και οι πάροχοι να μπορούν να εμπλακούν σε μια συζήτηση σχετική. Πέμπτο σημείο. Αξιοπιστία. Και εδώ είναι το θέμα, μπαίνει το θέμα της ευθύνη. Και εδώ πρέπει να υπάρχουν σαφεί κανόνε, γιατί αλλιώς ε, θα του δημιουργήσει από μόνη τη η αγορά. Η Volvo, α πούμε, ανακοίνωσε ο πρόεδρο τη ότι η αποφυγή δυστυχημάτων και τα σχετικά συστήματα ε, θα τα συμπεριλάβει στην ε, κατασκευή των νέων μοντέλων. Θα πρέπει ίσως βεβαίως να υπάρξει και ένα σχετικό νομικό πλαίσιο για το θέμα της ευθύνης, ε, του κατασκευαστού, του εμπορικού αντιπροσώπου. Και τέλος, το θέμα των υποδομών. Δεν θα πρέπει να το ξεχνούμε. Και εδώ ε, είπα και άλλες χώρες ε, ευρωπαϊκές έχουν, έχουν προχωρήσει πολύ μπροστά πρέπει να δούμε τι γίνεται με το car-to-car communication, με το car-to-infrastructure communication, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε θετικά. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους σας. Ε, έχουμε μια πίεση χρόνου πάλι, οπότε εγώ δυστυχώς θα πρέπει να φύγω. Ο κύριος Κόχ ο κύριος Αντιπρόεδρος, θα αναλάβει για να προχωρήσετε στην, ε, στις ερωτήσεις και τις απαντήσεις. Ευχαριστώ όλους τους συμμετέχοντες που ήσασταν εδώ σήμερα. Ευχαριστώ που εμπλουτίσατε τη συζήτησή μας με τις παρεμβάσεις σας. Και τώρα δίνω την προεδρία στον κύριο Κόχ. Äh, Τρεις ερωτήσεις βλέπω. Ο κύριος Λούγκριν έχει το λόγο πρώτος. Thank you, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τώρα ταχύτητας στη Γερμανία. Πριν από 1,5 χρόνο πήγα σε φορτηγό και ήμουν πριν από 10 χρόνια και κυκλοφόρησα για πάρα πολλές ώρες στους γερμανικούς αυτοκινητοδρόμους και έβλεπα εκεί τις BMW, τις Porsche και όλα τα άλλα μεγάλα αυτοκίνητα και έβλεπα Μα γιατί να πληρώνει κανεί τόσα χρήματα για να έχει ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Για το μέσο όρος ταχύτητας είναι όσο μπορεί να φτάσει ένα Fiat Panda. Οπότε γιατί να μην αγοράσει Fiat Panda αφού τόσο μπορείς να τρέξεις. Σε μερικέ περιπτώσεις το βράδυ μπορείς να χρησιμοποιήσεις βέβαια περισσότερη ισχύ αλλά ο μέσος όρος ταχύτητας είναι χαμηλός. Τώρα όσον αφορά τα λιγότερο βαριά οχήματα, είτε στους γερμανικούς αυτοκινητοδρόμους, είτε στους ευρωπαϊκούς, ο μόνος λόγος, το μόνο που θα μπορούσε να βοηθήσει θα ήταν τα μέγα τραξ που θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν τρία ευρωπαϊκά μοντέλα φορτηγών και τότε θα έχει νόημα. Για να πάει κανείς από τη Βόρεια Γερμανία ως το Μόναχο με το Omega Track, φυσικά κάποια στιγμή θα έπρεπε να το διαρρέσει πάλι σε τρία κομμάτια για να φτάσει στους ανθρώπους που έπρεπε να προμηθεύσεις. Το θέμα του ελέγχου ταχύτητας λοιπόν είναι το πιο περίεργο που άκουσα σήμερα. Όταν κάποιος με μεγάλη ταχύτητα τρέχει στους δρόμους, ο κόσμος που το βλέπει, τι νομίζετε ότι σκέφτεται, ότι α, πω, αυτός κινδυνεύει ή έχει πιει και γι' αυτό τρέχει. Όχι. Ο κόσμος ξέρει πολύ καλά ότι δεν πρέπει κανείς να πίνει και να οδηγεί. Και κανείς δεν θα συνδέσει την ταχύτητα του Σεμπάστιαν Πέκελ με τον Τζόνι Βόκερ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, ε, Ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να αναφερθώ στο ποτό, στο αλκοόλ. Φυσικά, εδώ μιλάμε για αλλαγή στη συμπεριφορά των οδηγών. Στην ε, Σουηδία, ευτυχώς, η κατανάλωση αλκοόλ έχει μειωθεί κατά πολύ. Έχουμε το λιγότερο από τα τελευταία 50 χρόνια. παρά τις διαφημίσεις όσων πουλούν αλκοόλ. Αντιστέκεται ο κόσμος. Θέλω όμως να ε, μιλήσω για αυτά τα alcohol logs. Στην αρχή αντέδρασε ο κόσμος και εγώ και είπα βεβαίως πρέπει να υπάρχει αυτός ο αποκλεισμός. Ήτανε σημαντικό λοιπόν για πάρα πολύ κόσμο για λόγους ασφάλειας και πολλές εταιρείες συμφώνησαν και η τεχνολογία βελτιώνεται όσο περνάει ο καιρός. Εντοπίζεται πιο εύκολα το κατά πόσο έχεις αλκοόλ στον οργανισμό σου. Όμως, τι γίνεται με την ομοθεσία. Γιατί να μην μπορεί να είναι υποχρεωτική αυτή, αυτός ο μηχανισμός από την ομοθεσία. Ευχαριστώ. Ε, έχω γράψει και εγώ το όνομά μου στον κατάλογο. να σας περιγράψω κάτι. Είμαι πίσω από ένα αυτοκίνητο, πατάει λίγο το φρένο, καταλαβαίνω εγώ ότι πρέπει και εγώ να πατήσω φρένο, δυστυχώς δεν ξέρω πόσο το μπροστινό αυτοκίνητο φρενάρει. Εντάξει, δεν χρειάζεται να έχω ένα φωτάκι που θα μου λέει ότι α, πρέπει και εσύ να πατήσεις λίγο φρένο, ε, γιατί ο μπροστινός ε, φρενάρει λίγο. Φρενάρω λοιπόν και εγώ λίγο. Αν φτάσω τη διάβαση των πεζών. Ωστόσο, δεν ξέρω αν με είδε αυτός που έρχεται με το φορτηγό. Ε, μήπως θα πρέπει ένα φωτάκι να ανάβει και να λέει ότι «Α, μπορείς να φύγεις τώρα». Ε, σε, κάποιες, ε, σε, κάποια, ε, σε κάποιους δρόμους μπορεί να γίνεται αυτό. θα μπορούσαμε ίσως να αποφύγουμε τέτοια είδου ατυχήματα. Δεν θα μπορούσαμε να σκεφτούμε κάτι παρόμοιο. Ναι, να πω ότι θα ξεκινήσουμε με την ίδια σειρά που ακούσαμε τις ε, παρουσιάσεις και θα έχουμε ένα μισή λεπτό για τον κάθε μιλητή για να απαντήσει. Sorry, ε, Mr. Van der Kamp. <laughs> Ο κύριος Van δεν σας έχω στην κατάλογο μου. Ναι, άργησα να ζητήσω το λόγο, ναι. Είμαι εδώ όλο το απόγευμα και ακούω και παρακολουθώ. Και όλα αυτά που λέτε είναι πολύ ενδιαφέροντα. Όμως έχω δύο ερωτήσεις. Και όχι τόσο πολύ για αυτό το πάνελ, ίσως περισσότερο για σας, κυρία μου, και για το προσωπικό εδώ. Οι 22.000 θάνατοι στους δρόμους έχουν αναλυθεί. Θέλω να πω πρόκειται για φορτηγά, πρόκειται για ιδιωτικά, ταχύ δηλαδή, πρόκειται για σκούτερ, για μηχανάκια, για πεζούς. Πολύ θα ήθελα να έχω περισσότερα στοιχεία. 22.000 νεκροί, τι είναι. Μια ανάλυση. Και δεύτερον, εδώ ήρθα για να ακούσω ένα πολύ δύσκολο θέμα, το οικονομικό κόστος από τους τραυματίες. Τελικά δεν άκουσα τίποτα γι' αυτό, ίσως έκανα λάθος. Μερικές φορές σκέφτομαι οι Ευρωπαίοι μπορεί να μην πίνουν πολύ, να μην τρέχουν πολύ, όμως το πορτοφόλι τους τους νοιάζει. Γι' αυτό ρωτάω, ποιο είναι το οικονομικό κόστος των βαριά τραυματισμένων για την κοινωνία, για τα κράτη μας. Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσετε εσείς. Ναι. Το πρόβλημα είναι όταν μεγαλώνουν οι υποδομές και αυτό σημαίνει μεγαλύτερη ταχύτητα. Το λέει και το και η TCS, το Συμβούλιο Δικής Ασφάλειας στην ιστοσελίδα τους. Και στη Γαλλία έχουν υπάρξει σχετικές εξελίξεις. Αυξήθηκε το, το όριο ταχύτητας, αυξήθηκαν και τα αυξήθηκαν όχι κατά ανάγκη τα ατυχήματα, αλλά αυξήθηκαν οι θάνατοι από ατυχήματα. Πολύ σημαντικά, λόγω της υψηλής ταχύτητας. Οπότε το όριο ταχύτητας είναι πολύ σημαντικό. Στη Γερμανία υπάρχουν πάρα πολλά Υπάρχει πολύ μεγάλη κυκλοφορία και συμφόρηση. μιλάμε για 160-180 ε, χιλιόμετρα με τα οποία μπορεί να τρέχει ένα αυτοκίνητο και ξαφνικά πρέπει να φρενάρει γιατί μπροστά του υπάρχει ένα φορτηγό και πρέπει να κατέβει στα 80. Ε, Βεβαίω όταν ένα μποτιλιάρισμα δεν ε, προχωράει αναρωτιέται κανένα τι γίνεται κυρίως όταν η κυκλοφορία είναι πάρα πολύ πυκνή. Τώρα για τα mega trucks, Ε, Προφανώ είναι πολύ πιο ασφαλέ ε, το ε, φορτηγό όταν το κοντέινερ του τουλάχιστον ή και το ίδιο έχει μεταφερθεί στον ε, σιδηρόδρομο. Νομίζω αυτό ήταν ένα στόχο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η μετάβαση στο, και η πρόθεση αυτή, η μετάβαση στον σιδηρόδρομο. Για την ασφάλεια τώρα την οδική, η VCD έχει κάνει έναν έλεγχο για τι διάφορε πόλει ε, οι θάνατοι καταμετρώνται και οι τραυματίες επίσης και αξιολογούνται για τις διάφορες πόλεις και υπάρχει και μια κατάταξη ας πούμε των ε, πόλεων. Ε, ίσως αυτό θα μπορούσαμε να το κάνουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ανά πόλη ή ανά χώρα και ανά ατυχήματα. Ευχαριστώ. Okay. Um, so Λοιπόν, ε, ρωτήθηκε ποιος ε, θα συσχετήσει τη Φόρμουλα 1 και το αλκοόλ στην οδήγηση. Κάποιοι θα το συσχετήσουν. Ε, βέβαια ταυτόχρονα είναι και ευθύνη των ατόμων. Αλλά έχουν φυσικά και οι κυβερνήσεις ένα καθήκον να μεριμνούν για τους πολίτες τους. Γι' αυτό έχουμε και την νομοθεσία. Εγώ αυτό προσπαθώ να πω είναι ότι έχουμε πρόβλημα όταν η βιομηχανία των ενοπνευματοδών υποστηρίζει το άριστο εξαιρετικό έργο της ETSC. Δηλαδή ε, ε, αυτή την πολιτική κατά της χρυσαλκόλ πριν την οδήγηση, αλλά ταυτόχρονα σαμποτάρει τις κοτσέζικες ε, αρχές όταν πάνε να εισάγουν ελάχιστη τιμή. Οπότε από τη μία υποστηρίζουν το έργο αυτό που έχω στα χέρια μου και από την άλλη είναι χορηγή μιας δραστηριότητα που δημιουργεί ένα σχετισμό μεταξύ του αλκοόλ και της οδηγήση. και ειδικότερα της γρήγορης οδηγήση. αγωνιστικού τύπου. Ευχαριστώ. Κατσίου. Μία ερώτηση όσον αφορά τα συστήματα κινητοποίησης του οχήματος, τα interlock. Οι οδηγοί μας, ξέρετε, χρησιμοποιούν ε, τα αυτοκίνητα ως ε, μέσα πραγματικής κινητικότητας ε, πατάνε ένα κουμπί, ξεκινούν τα αυτοκίνητα αυτόματα.